9 η ώρα, επομένως αρχίζουμε. Κηρύττω την έναρξη. Έχουμε μία ημερήσια διάταξη. Το σημείο 8 δεν θα το εξετάσουμε σήμερα, αλλά θα μεταφερθεί στην επόμενη συνεδρίασή μας. Πρόκειται για τα θέματα πολιτισμού στην υπηρεσία εξωτερικών ε, δράσεων. Αλλά επειδή ο προπολογισμό δεν έχει εγκριθεί και δεν έχουμε καθόλου χρήματα για την υπηρεσία εξωτερική δράση, έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε και λίγο καλύτερα για αυτά που θέλουμε να αποφασίσουμε στον τομέα αυτό. Επομένω, για πρώτη φορά το Δεκέμβριο θα εξετάσουμε αυτή την έκθεση για τον πολιτισμό και θα συζητήσουμε Πρόκειται για την έκθεση ΣΑΚΕ. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει για την ημερήσια διάταξη, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. Ε, όπως ξέρετε, μεταδίδεται και στην τηλεόραση, ή τουλάχιστον στο ίντερνετ, συνεδρίασή μας. Έχουμε μετάφραση σε όλες τις γλώσσες, εκτός από τα εστονικά, τα λετονικά, τα μαλτέζικα και τα σουηδικά. Όλες οι άλλες γλώσσες παίζουν στο γήπεδο. <clears throat> Επίσης, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι έχουμε εδώ τον Πολωνό Υπουργό Αθλητισμού εδώ μαζί μας για την ακρόαση που θα κάνουμε σε λίγο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει και το Συμβούλιο των Υπουργών να ασχοληθεί με τα θέματα του αθλητισμού. Είναι πολύ καλό λοιπόν να έχουμε κάποιον ο οποίος όχι μόνο είναι υπουργό, αλλά είναι υπουργό από τη χώρα που θα αναλάβει τη σκητάλη της Προεδρίας και είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις του Υπουργού Αθλητισμού και θέλω σας παρακαλέσω να κάνετε κάτι που δεν έχετε κάνει μέχρι τώρα, να ψηφίσετε για το βραβείο Λουξ. Σας παρακαλώ, εκ βάθους καρδίας, όχι μόνο εσείς οι ίδιοι, αλλά να πείσετε άλλους πέντε συναδέλφους σας τουλάχιστον να ψηφίσουν για το βραβείο αυτό. Για να μπορέσει αυτό το βραβείο <clears throat> να έχει συνέχεια στο χρόνο, αυτό θα εξασφαλιστεί μονάχα αν δείξουμε εμεί ενδιαφέρον. Αν εμεί δεν ψηφίζουμε, αν έχουμε προβλήματα, ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι κατά το βραβείο αυτού Λουξ, θα στραφούν εναντίον αυτού του βραβείου. Εγώ ήμουν χθε την ε, ήμουνα το Σάββατο, το, την Κυριακή στο Μόναχο και μετά στο Βερολίνο και είδα ότι υπήρχε πολύ ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά και για πρώτη φορά άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ιδέα τι ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασαν τη χαρά τους και το ενδιαφέρον τους για το γεγονός ότι εμείς προσπαθούμε με την ιδέα αυτή του βραβείου Λουξ να υποστηρίξουμε τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο και να δώσουμε ως τον μεγαλύτερη διάδοση στα πολιτιστικά αγαθά της Ευρώπης. Μπορεί να είναι σταγόν εν το ωκεανό, αλλά είναι σταγόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό σα παρακαλώ, όλοι οι παρόντε συνάδελφοι θα πρέπει να ψηφίσουν και να προσπαθήσουν να πείσουν τουλάχιστον πέντε συναδέλφου από το περιβάλλον του στο στενό για να ψηφίσουν και αυτοί. Εντάξει. Μη με απογοητεύσετε λοιπόν. Και εξάλλου υποστηρίζετε με τον τρόπο αυτό κάτι το οποίο είναι θαυμάσιο. Ψηφίστε λοιπόν ε, νομίζω ότι μόνο ένας από εσάς έχει... Δεν έχει ψηφίσει. Δεν έχει ψηφίσει. Α, ολότερα έχει ψηφίσει. Εντάξει, είναι αθώος. Ωραία. Αυτά για τις ανακοινώσεις. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο θέλω να σας πω. Την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη του Στρασβούργου, θα έχουμε μια παράσταση θεατρική στο Κοινοβούλιο. Το Jean Théâtre Public στο Στρασβούργο θα κάνει μια παρουσίαση στις ε, μία η ώρα στην καφετέρια. Πρόκειται για νέους φοιτητές οι οποίοι θα μας ε, κάνουν αυτή τη μεγάλη χαρά να έρθουν στο Κοινοβούλιο την Τρίτη το μεσημέρι και να κάνουν μια παράσταση. Και φυσικά θα σας, μια, θα σας στείλουμε μια πρόσκληση. Σας παρακαλώ να έρθετε λοιπόν και να είσαστε εκεί για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και να του χειροκροτήσετε. Λοιπόν, πρώτο που είμαι στην ημέρα διάταξη, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε ένα άτομο το οποίο είναι μαζί μας για τελευταία φορά, στην τελευταία, μας, τελευταία συνεδρίαση μαζί μας. Χάνουμε σημαντικές δυνάμεις, ε, δεν χάνεται, πηγαίνει σε μια υψηλότερη θέση, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει και μια εναλλαγή του προσωπικού, οι άνθρωποι να μην μένουν πάντα παγιωμένοι σε μια θέση. Λοιπόν, Γιούργεν, λυπάμαι, αλλά είχαν τόσα πολλά για την Επιτροπή μας και για τον αθλητισμό, που να μην μπορώ να ξέρω αν θα είναι δυνατόν να σε αντικαταστήσουμε. Θα μας λείψεις όμως γιατί έχεις κάνει μια εξαιρετική εργασία στην Επιτροπή μας. Πάρα πολλέ συζητήσει που κάναμε δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα στην Επιτροπή μα, ακόμα και την εποχή που δεν ήμουνα πρόεδρο τη Επιτροπή και νομίζω ότι πάρα πολλά μέλη τη Επιτροπή μα συμμερίζονται την ευγνωμοσύνη μου για τον Γιούργεν και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το χειροκροτήσουμε. Ωραία, δουλειά. Έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική ψηφοφορία. Ξέρω ότι η Ελβετία είναι ουσιαστικά κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει σε πάρα πολλά προγράμματα, συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας στο Youth for Action και στο πρόγραμμα διαβίου μάθησης. Όλα αυτά δεν κοστίζουν ουσιαστικά σε μας. Έχουμε ανοιχτές ε, ε, πόρτες για όλους. Επομένω, όλα αυτά υποστηρίζονται από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη δική μα πλευρά, αλλά η Ελβετία θα πρέπει να τα υποστηρίξει και με το δικό τη προπολογισμό και πρέπει να ψηφίσουμε βάσει του άρθρου 182 παράγραφος 6 της Συνθήκης της Λισαβόνας θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε στο Συμβούλιο για το κατά πόσο συμφωνούμε με τη συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους Ελβετούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό και ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει την Ελβετία να βρει καλύτερα το δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπαμε είναι με το ένα πόδι μέσα, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα υπάρξει και μια απόφαση σε μορφή δημοψηφίσματος στην Ελβετία για να γίνουν μέλη. Έχουμε λοιπόν μόνο μία ψηφοφορία να κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε κάρτες ε, ψηφοφορίας. Ποιος υποστηρίζει την συμμετοχή της Ελβετίας σε αυτά τα προγράμματα. Κατά. Αποχές. Αποχές, κανείς αποχές. Ομόφωνα δεκτή. Χαιρόμαστε λοιπόν για τη συμμετοχή της Ελβετίας σε αυτό το πρόγραμμα. So, Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στη δημόσια ακρόαση για τη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική αθλητισμού. Ξέρετε όλοι ότι έχουμε, έχει περατωθεί η μελέτη που έχουμε ζητήσει να γίνει για τα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής αθλητισμού μέσα στα πλαίσια της νέας συνθήκης της Λισαβόνας και φυσικά αυτή η μελέτη βασίζεται σε μια πραγματικότητα ότι δεν υπάρχουν μεν πολλές πραγματικές δυνατότητες, αλλά έχουμε πολλές φιλοδοξίες βάσει του, της συνθήκης Λισαβόνας. Η ιδέα της παιδεία μέσω του αθλητισμού ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία με πολύ καλά αποτελέσματα, στι πρακτικέ εμπειρίε που συλλέξαμε και όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Επίση, δώσαμε και την άποψή μα για την Λευκή Βιβλία της Κομισιόν. Ο τότε συνάδελφό μα κ. Μαυρομάτη εργάστηκε για τα θέματα αυτά. Έχουμε και μια γραμμή του προπολογισμού για την υποστήριξη μέτρων στον τομέα του αθλητισμού κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι είδαμε και το είδαμε και στην τελευταία μας ε, συνεδρίαση όταν παρουσιάστηκε αυτή η μελέτη ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιδιαίτερα το άρθρο της Συνθήκης Λισαβόνας για τα θέματα όταν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και άλλα μέτρα. Στις αρχές του καλοκαιριού κάναμε μια ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν ναι, για το θέμα των player agents, των manager των παιδιών, των παικτών κύριος Χόλγκερ ίσως μπορεί να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Με το άρθρο της συνθήκης της Λισαβόνας, όπως ελέγχθη, έχουν ξεκινήσει πολλές προσδοκίες, αλλά οι οποίες έχουν διαψευστεί σε μεγάλο βαθμό. Η Επίτροπος κυρία Βασιλείου στην τελευταία μας συνεδρίαση μας δήλωσε ότι μέχρι, το επόμενο, μέχρι, την τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, μέχρι το, τον επόμενο χρόνο πολιετών ε, προοπτικών δεν θα μπορέσουμε να έχουμε σημαντικά νέα προγράμματα στον αθλητισμό. Αυτό βέβαια ήταν απογοητευτικό. Πρέπει όμως, να, εφόσον δεν θα έχουμε κάτι καινούριο μέχρι το 2013, να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα μέσα που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας. Πάντως, μετά από το 2013 θα πρέπει να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε. Γιατί αν δεν τα κάνουμε αυτό μπορεί να μην υπάρχουν αυτά τα προγράμματα τότε. Και πρέπει να δούμε τώρα πού βρίσκονται τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα θέματα του αθλητισμού στον προϋπολογισμό. Ελπίζω ότι δεν θέλουν τα περισσότερα, κράματα, τα περισσότερα κράτη-μέλη να υποβιβάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην δεύτερη κατηγορία, δηλαδή σε μια ένωση κρατών που είναι απλώς μια εμπορική ένωση. Πρέπει να αγωνιστούμε λοιπόν για όλα αυτά τα πολιτιστικά προγράμματα, όπως και για τα προγράμματα του αθλητισμού. Και για αυτό το λόγο σας παρακαλώ να σκεφτείτε συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού. Υπάρχει λοιπόν μια μικρή αμυδρά ελπίδα ότι κάτι θα προχωρήσει και ότι θα υπάρξει και μια λήψη απόφασης σε επίπεδο λιπτών απόφασης για να έχουμε μια πιο πραγματική πολιτική στα θέματα του αθλητισμού. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα μπορούμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση η οποία θα μπορέσει να δώσει και κάποιο έναυσμα σε περαιτέρω ενέργειες από το Συμβουλίο των Υπουργών. Είναι η σωστή μέρα λοιπόν για μια τέτοια ακρόαση. Ευχαιρετίζω όλους τους εμπειρογνώμονε μας. Έχουμε φυσικά τον Γκρέγορη Πόλκερ από την Κομισιόν, από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση που ασχολείται με τα θέματα αθλητισμού και χαιρόμαστε ότι ο, ο Πάτρικ Κέι είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή, από την UEFA έχουμε το William Γκαγιάρο, ο οποίος είναι σύμβουλο του Μισελ Πλατινί. Έχουμε επίσης από το Διεθνή Φορέα το, ε, για τον Αθλητισμό και την Κουλτούρα, το Μόρκεν Κίρκεβι. Και έχουμε και τον καθηγητή για το, για το Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο, τον Μισελ Κολούτσι. Την κυρία Μισελ Κολούτσι, θου κυρία φυλακή το στόματί μου. Γυναίκα είναι, ναι, όχι άντρας. Συγγνώμη Μισελ, συγγνώμη Μισελ. Στα γαλλικά είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανεί άντρε και γυναίκε όταν λέγονται Μισελ. Αν νόμιζα ότι λέγονταν Μικέλε. Α, Μικέλε. Πολύ ωραία. Ο Μικέλε Κολούτσι. Χαίρομαι λοιπόν που είσαστε όλοι εδώ πέρα και προτείνω την εξή διαδικασία. Να ακούσουμε καταρχήν τον κύριο Πάλγκερ από την Κομισιόν και μετά θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες να μας δώσουν τις απόψεις τους και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και σχόλια των συναδέλφων και θα δώσουμε μετά στην Κομισιόν την ευκαιρία να απαντήσουν και θα ακούσουμε και τη Βελική Προεδρία γιατί θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις απόψεις μας στην, στην Σύνοδο των Υπουργών για τα θέματα πολιτισμού. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το σφυρί μου αν ξεπεράσετε το χρόνο σας, αλλά σας παρακαλώ να μην χρειαστώ να το κάνω αυτό. Κύριε Πόλγερ, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Να σας πω πως είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι ξανά στην Επιτροπή σας με τα νέα μου καθήκοντα ως Διευθυντής Νεολαίας και Άθλησης. Είμαστε σε μια περίοδο μετά την Λισαβόνα. Έχουμε ειδική συγκεκριμένη αρμοδιότητα για τον αθλητισμό συμπληρωματική θα έλεγα μέσω του ευρωπαϊκού επίπεδου πρόθεσης του αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 165 μπορούμε να φέρουμε μια προστιθέμενη αξία στον τομέα του αθλητισμού και σχετικές φιλοδοξίες ένωσης στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 και να προωθήσουμε καλύτερα τον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Ως πρώτο βήμα αυτών των νέων διατάξεων η Κομισιόν Σύντομα θα ευθύσει μια ανακοίνωση με προτάσεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό που θα περιέχει συγκεκριμένα μέτρα και θα απευθύνεται στο Συμβούλιο και βεβαίως στο Κοινοβούλιο. Ε, στην ουσία τώρα της ανακοίνωσης θα τονίζει τη συνεισφορά του αθλητισμού και της ενεργητικής ε, αναψυχής ε, στην καταπολέμηση της ανεργίας, την διαρκή απασχόληση και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Βασική ιδέα είναι να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση με συγκεκριμένες δράσεις, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αθλητισμού. Στην εφαρμογή της βεβαίως θα απαιτήσει ενισχυμένη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως το αθλητικό κίνημα η ανακοίνωση θα βασιστεί στη Λευκή Βίβλο του 2007, το σχέδιο δράσης Pierre de Coubertin. Οι συγκεκριμένες δράσεις που θα υποβάλλουμε αντικατοπτρίζουν κυρίως τις ιδέες ε, που εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι και θα σεβαστούν βέβαια πλήρως την συνθήκη. Δηλαδή, το νέο αυτό θεματολόγιο θα υποστηρίζει την δράση στο εθνικό επίπεδο σε τομεί όπου η Ένωση μπορεί να προσθέσει κάποια αξία. Αυτό θα γίνει με διάφορους τρόπους, τους οποίους θα απαριθμίσω εντάχει. Να αφαιρθούμε σε διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στην Ευρώπη, να συνεισφέρουμε ως γενικότερους στόχους στρατηγικής 2020, να στηρίξουμε τις δράσεις των κρατών μελών και να τις ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε το πώς ε, θα αναπτυχθεί η γνώση στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων, το να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, να προωθήσουμε τη δημιουργία δικτύων στον ευρωπαϊκό αθλητισμό και να προωθηθεί η γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα του αθλητισμού. Βεβαίως, ε, θα καλυφθούν τομείς συγκεκριμένα όπως η κοινωνική συνοχή στον αθλητισμό μέσω και τον αθλητισμό των αναπήρων, ε, τις γυναίκες στον αθλητισμό, τους μετανάστες και τις μειονότητες. Το θέμα της διπλής καριέρας για νέους αθλητές υψηλού επίπεδου και το πώς θα συμπεριληφθούν στα εθνικά συστήματα προσόντων και τα αθλητικά προσόντα. Τρίτον, η, φυσική, η σωματική δραστηριότητα που ενισχύει την υγεία. Κάτι το οποίο παίζει ζωτικό ρόλο για την υγεία του εργαζόμενου πληθυσμού και άρα και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Την καταπολέμηση του ντόπινγκ και την ε, σωματική και ηθική ακαιρεότητα των αθλητών την καταπολέμηση κάθε είδους βίας ε, και μη ανεκτικότητας από πλευράς των θεατών, την αηφόρο ε, χρηματοδότηση του αθλητισμού μέσω ζητημάτων όπως η πνευματική ιδιοκτησία, το στίχημα και την κοινή πώληση δικαιωμάτων στα ΜΜΕ στήριξη των δομών αυτών μέσω ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων, πρόθεση της ορθής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, κανόνων για τους μεταγραφές ε, και βεβαίως στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο και επειδή του χρόνου είναι το ευρωπαϊκό έντος εθελοντισμού, ο εθελοντισμός στον αθλητισμό. Οπότε η ανακοίνωση θα καλύψει ε, τεράστιους τομείς αλλά τους άλλως ο αθλητισμός καλύπτει ένα τεράστιο τομέα και αναμένουμε το τι θα μας πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες με βάση αυτή την ανακοίνωση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Μπάγκα. Ο Πάτρικ Χίκε για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που παίρνω μέρος σε αυτήν την ακρόαση για την μελλοντική αθλητική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομιλώ σαν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών. Είμαι επίσης πρόεδρος της, ε, του, Ολυμπιακού Συμβουλίου της Ιρλανδίας. Ε, από ε, νέος ασχολούμαι με τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, από το βασικό επίπεδο, το απόλυτα ερασιτεχνικό μέχρι το επαγγελματικό και νομίζω ότι πρέπει να δούμε το θέμα του αθλητισμού με δύο συμπληρωματικούς τρόπους που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω ποιες είναι οι Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές. Δημιουργήθηκαν το 1975. Είναι ένας πανευρωπαϊκός αθλητικός οργανισμός που εκπροσωπεί σήμερα 49 Ολυμπιακές επιτροπούμε το Ολυμπιακό κίνημα στην Ευρώπη, οργανώνουμε τις δικές μας αθλητικές συναντήσεις, το φεστιβάλ, το αθλητικό, τους ε, χειμερινούς αλλά και τους θερινούς αγώνες για τους νέους από τις 49 χώρες και θεωρείται ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οικονομική βοήθεια που έδωσε στα, στους αγώνες ε, του 2009 στο Τάμπερε και που θα χρηματοδοτήσει τους αγώνες του Λίμπερετ στην ε, Τσεχία ε, την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος συνεργασίας ανάμεσα στο Ολυμπιακό κίνημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή μας από το Φεβράριο του 2009 έχει δημιουργήσει ένα βασικό γραφείο στην, μια αντένα μάλλον στις Βρυξέλλες, ενώ το κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στη Ρώμη. Εκπροσωπεί το γραφείο αυτό τα συμφέροντα των Ολυμπιακών Επιτροπών και άλλων 90 αθλητικών οργανισμών. Στόχος της αντιπροσωπείας αυτής είναι η σωστή εκπροσώπηση των συμμετεχόντων στα ευρωπαϊκά όργανα από την αρχή που δημιουργήθηκε. Στόχος είναι η συνεισφορά σε μια καλύτερη αθλητική πολιτική η οποία εξελίσσεται εδώ και 10 χρόνια περίπου. Η αναφορά στον αθλητισμό στη συνθήκη της Λισαβόνας και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα είναι αλήθεια ότι εμείς μόνο το Δεκέμβριο του 9 ασχοληθήκαμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας Είχαμε βέβαια το 2003 και 2004 ασχοληθεί με αντίστοιχα θέματα στα πλαίσια της συνέλευσης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Τότε η συμπερίληψη του αθλητισμού είχε υποστηριχθεί από τις αθλητικές οργανώσεις. Υποστηρίξαμε επίσης και την αναφορά στη νέα συνθήκη της Λισαβόνας όταν έγινε δεκτή από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το 2007 Προσπαθούμε να πετύχουμε συγκεκριμένες προσδοκίες που έχουν τα μέλη μας. Θυμάμαι μια εκστρατεία η οποία λεγόταν Ευρωπαϊκή Ένωση και Αθλητισμός, η επίτευξη και ολοκλήρωση όλων των προσδοκιών. Πράγματι είχαν δημιουργηθεί στο αθλητικό και στο ολυμπιακό κίνημα πολλές προσδοκίες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσουμε να διαμορφωθεί καλύτερα η νέα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αθλητικό τομέα. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2008 με το Φόρουμ για τον Αθλητισμό θα βοηθήσουμε και βοηθήσαμε να αντιμετωπίσει τις κοινέ προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το παράνομο στίχημα, η εκπαίδευση και προστασία των νέων αθλητών, τα αθλητικά σχολεία κτλ. Διατηρώντας βέβαια πάντα τον ειδικό χαρακτήρα της αθλητικής δραστηριότητας. Είχαμε πολλές συναντήσεις το 2009 με τον Επίτροπο Φίγκελ, είχαμε μια εξαιρετική σχέση μαζί του και μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας συντονίσαμε την κοινή μας θέση στα πλαίσια του Ολυμπιακού κινήματος για την εφαρμογή της νέας συνθήκης στους κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό. Οι προτάσεις μας έχουν κατατεθεί ε, στα κράτη-μέλη και στα ευρωπαϊκά όργανα στις αρχές του 2010. Τώρα για τη συνθήκη της Λισαβόνας και το Ολυμπιακό κίνημα. Να υπογραμμίσω ποια είναι τα βασικά στοιχεία ε, τα οποία εμείς προωθούμε τα ειδικά χαρακτηριστικά ε, του αθλητισμού και της αθλητικής δραστηριότητας πρέπει να είναι η βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον αθλητισμό. Η πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται στο παρελθόν από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τώρα πλέον τα ευρωπαϊκά όργανα ε, να μπορέσουν να ξεπεράσουν την απλή ξερή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομολογίας και να μπορέσουν να περάσουν και σε νομοθετικές δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού, δημιουργώντας μια νέα κοινοτική αρμοδιότητα. Θεωρούμε ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού έχουν μεγάλη αξία. Η δήλωση για τον αθλητισμό που προσαρτήθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2008 λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού πέραν των οικονομικών χαρακτηριστικών Ξέρω ότι πολλοί θεωρούν ότι αυτή η δήλωση δεν έχει νομικά δεσμευτικές επιπτώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δηλώσεις τέτοιες δίδουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλικό για σκέψη και υλικό για να προχωρήσουν στην εφαρμογή της νέας κοινοτική νομοθεσίας. Εμείς υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία και αυτονομία των αθλητικών ομοσπονδιών και το δικαίωμά τους να ορίσουν την οργανωτική τους ε, δομή. Νομίζω ότι η κοινή πολιτική θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη ε, των, ε, της σωστής εφαρμογής των διεθνών κανόνων για το fair play στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα και θα πρέπει να υπάρξει και περαιτέρω χρηματοδότηση των αθλητικών προγραμμάτων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανησυχώ για τι τελευταίε ανακοινώσει που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μου φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξε και ίσω να είναι και ένα μείζον βήμα προ τα πίσω. Το βασικό αθλητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κύρια πρωτοβουλία την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τον αθλητισμό. Όλοι, κοιτάξτε, δεν έχουμε πάρα πολλά λεπτά. Είχαμε 4 με 5 λεπτά. Δεν μπορώ να σας αφήσω άλλο χρόνο. Θα συνεχίσω. Ελπίζω το Συμβούλιο Υπουργών να πάρει μια σωστή απόφαση γύρω από το θέμα αυτό και να μην είναι φλιαρίες. Ο κύριος Γκαγιάρ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε στην Επιτροπή σας ε, εξ ονόματος της UEFA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομαδικών Αθλημάτων. Είναι παράδοξο όταν συζητάμε για την ευρωπαϊκή πολιτική αθλητισμού και ο αθλητισμός γίνεται για πρώτη φορά μια κοινοτική αρμοδιότητα να ξεχνάμε να πούμε ε, τα βασικά χαρακτηριστικά, να αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά της, του αθλητισμού ε, θα έλεγα στην Ευρώπη, το ευρωπαϊκό αθλητικό πρότυπο. Γιατί είναι σημαντικό το πρότυπο αυτό να αναγνωριστεί ε, και να θεωρηθεί κυρίαρχο από πλευρά των ευρωπαϊκών οργάνων. Η απάντηση είναι ταυτόχρονα απλή γιατί είναι ένα πρότυπο θα έλεγα αλληλέγγυο και αντιπροσωπευτικό για όλη την Ήπειρο αλλά και ιδιαίτερα περίπλοκο γιατί το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει στο εσωτερικό του όλες τις αποχρώσεις και όλες τις έφραστες ισορροπίες οι οποίες του προσδίδουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει το ευρωπαϊκό αθλητικό κίνημα. Αλληλέγγυο και αντιπροσωπευτικό είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Ο ευρωπαϊκός αθλητισμός είναι ένα σύνολο. Σχηματικά παρουσιάζεται σαν μια πυραμίδα της οποίας η βάση αποτελείται από εκατομμύρια αθλητών, αθλουμένων μάλλον τα διάφορα επίπεδα της πυραμίδας αυτής αντιπροσωπεύουν τα τοπικά επίπεδα, επαρχιακά, περιφερειακά και εθνικά επίπεδα όπου περιλαμβάνεται το ε, ερασιτεχνικό σπορ, τα, τα ερασιτεχνικά αθλήματα, τα παιδικά αθλήματα και όσο πιο ψηλά πηγαίνει κανείς αυτή την πυραμίδα τόσο πιο διαφοροποιείται, τόσο πιο εξειδικεύεται και οι αθλητικές δραστηριότητες και ο ανταγωνισμός αυξάνεται και, λιγότερο, και γίνεται λιγότερο κοινωνικός. Αεραστεχνικά χαρακτηριστικά αντικαθίστανται από τον επαγγελματισμό και το πάθος αντικαθίσταται από την καριέρα οι αθλητικές ομάδες ε, εντάσσονται σε ε, ομοσπονδίες, σε ενώσεις των οποίων οι διευθυντικές ε, επιτροπές εκλέγονται δημοκρατικά σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα ε, τα αθλήματα οι επαγγελματικές ενώσεις αντιπροσωπεύουν κάτω του 1% των αθλωμένων. Αλλά χάρη στην οικονομική αλληλεγγύη η οποία είναι το θεμέλιο του ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου αυτή η ελίτ, η ελαχιστοτάτη αλλά ιδιαίτερα ευημερούσα ε, χρηματοδοτή και διατηρεί εν ζωή, αν θέλετε, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ο επαγγελματικός τομέας τροφοδοτεί σε κάθε ομοσπονδία τις βασικές αθλητικές δραστηριότητες, είναι κάθε η λειτουργία του αλλά και οριζόντια. Σαν παράδειγμα στο ποδόσφαιρο η UEFA μοιράζει και ανακατανέμει τους πόρους της στις 53 ομοσπονδίες τις ποδοσφαιρικές όπου οι πιο πλούσιες ουσιαστικά χρηματοδοτούν τις φτωχότερες το σύστημα επιτρέπει επίσης και την κοινότητα και την κινητικότητα, συγγνώμη, πέραν της κατανομής ανάμεσα σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές. Προσπαθούμε να προωθήσουμε ε, ε, την, ε, τις αλλαγές στην ιεραρχία όλων των επιπέδων της πυραμίδας και στο ποδόσφαιρο αλλά και στα υπόλοιπα αθλητικά αθλήματα δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι μόνο σε μία κατηγορία όπως το έχει υπογραμμίσει ο πρόεδρος της UEFA, ο Μισελ Πλατινί, στις αρχές της χρονιάς εδώ στις Βρυξέλλες, το ευρωπαϊκό αθλητικό πρότυπο βασίζεται σαν σύνολο στην ιεραρχική κινητικότητα και την αλληλεγγύη. Είναι κάτι το μοναδικό και βαθύτατα ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι οι επαγγελματικές αθλητικές δραστηριότητες μερικές φορές αναζητεί τη σωτηρία τους σε μια θα έλεγα διαφυγή προς το μέλλον σε οικονομικό επίπεδο που δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό θα πρέπει να αντιστραφεί γιατί απειλεί το κοινωνικό μας ιστό και την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και το μέλλον της νιώτης στην Ευρώπη. Η Επιτροπή σας έχει μια ευκαιρία η οποία ίσως να μην επαναληφθεί να πλαισιώσει το ευρωπαϊκό αθλητικό πρότυπο και να το καταστήσει βασικό θεμέλιο των πολιτιστικών αξιών της Υπήρους μας. Ελπίζω να μην χάσετε την ευκαιρία αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει και η πρόεδρος ΠΑΚ <clears throat> και ιδίω γιατί παραμείνατε μέσα στα πλαίσια του αγωνιστικού χώρου, δηλαδή των πέντε λεπτών. Και ήταν πολύ καλό και το περιεχόμενο εξάλλου. Χωρίς μικρόφωνο η Πρόεδρος. Διεθνής Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξέρω ότι έχω μονάχα πέντε λεπτά, γι' αυτό θα πάω κατευθείαν στο ψητό το άρθρο της συνθήκης της Λισαβόνας που έχει προσθεθεί για τα θέματα του αθλητισμού, αυτό είναι μια έμπνευση για να έχουμε πραγματικά μια πιο εμπεριστατωμένη δραστηριότητα στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού και είναι η βάση για όλους τους λήπτες αποφάσεων. Δεν ανοίγει την πόρτα μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για φιλοδοξίες, πολιτικές <clears throat> φιλοδοξίες και αποφάσεις που μπορούν να έχουν μεγάλη επίπτωση στην κουλτούρα και στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Στι δύο τελευταίε δεκαετίες η Ευρώπη έχει αναπτυχθεί, έχει εξελιχθεί και το ίδιο και οι πολίτε της έχουν νέε προοπτικέ, νέε απαιτήσει για τα σπορ και τη σωματική δραστηριότητα. Με τη νέα συνθήκη θα έχουμε μια πολύ καλή πλατφόρμα για να αναπτύξουμε τη σωματική άσκηση και τον αθλητισμό, αλλά είναι απαραίτητο να ξεπεράσουμε ορισμένου μύθου και πεπαλαιωμένα υποδείγματα σε σχέση με τον αθλητισμό. Θα πρέπει να βασιστούμε στα στοιχεία και στη γνώση. Με τη σημερινή συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε το σωστό επίπεδο <clears throat> συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να δημιουργήσει ένα όραμα το οποίο θα συναθρήσει τους εμπλεκομένους από διάφορους τομείς και όχι μόνο από τον περιορισμένο τομέα του αθλητισμού αυτόν καθεαυτό. <clears throat> Έτσι ο αθλητισμός μπορεί να πλησιάσει και να αγγίξει περισσότερους πολίτες και να χρησιμοποιήσει και περισσότερους πόρους. Αυτό το κοινό όραμά μας λοιπόν σημαίνει ότι 100 εκατομμύρια παραπάνω πολίτες Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ενεργοί στη σωματική άσκηση και τον αθλητισμό μέχρι το 2020. Πρωτού όμω περάσω σε αυτό, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα για τη σωματική άσκηση και τον αθλητισμό στην Ευρώπη σήμερα. 200 εκατομμύρια ή 40% όλων των Ευρωπαίων θεωρούν ότι ασκούνται και ότι κάνουν σπορ σε τακτική βάση. 34% όμως όλων των Ευρωπαίων είναι αδρανείς στον τομέα αυτό ή ασκούνται πάρα πολύ σπάνια. Υπάρχουν 70 εκατομμύρια σε αθλητικούς ομίλους, αλλά είναι και 130 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίων που ασκούνται αθλητικά σε εκτός των ομίλων. Οι προτιμήσεις είναι η άσκηση στα πάρκα και στη φύση ένα 30% σε ομάδες αθλητικούς, αθλητικές και ενώσεις και πρέπει να τονίσουμε ότι ακόμα και αν το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ ορατό άθλημα οι Ευρωπαίοι προτιμούν να περπατούν, να κολυμπούν, να κάνουν ποδήλατο και να κάνουν άσκηση στο γυμναστήριο. <clears throat> Γιατί θέλουν να βελτιώσουν και τη σωματική τους υγεία και να διασκεδάσουν επίση. Αυτά είναι τα πράγματα που ενδιαφέρουν του Ευρωπαίου σήμερα. Επανέρχομαι τώρα σε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένω. Γιατί ακούσαμε για το μοντέλο πυραμίδα. <clears throat> Μας έχει παρουσιαστεί πολλές φορές και θα έπρεπε να καταδεικνύει πώς λειτουργεί ο αθλητισμός σήμερα στην Ευρώπη. Αλλά αυτό το υπόδειγμα πυραμίδα δεν καταδεικνύει την πραγματικότητα στον αθλητικό τομέα. Γιατί η βάση της πυραμίδας έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αναφέρθηκε το θέμα της ε, ε, οικονομικής αλληλεγγύης και του μάρκετινγκ. Και εδώ θέλω να σταθώ κάποια στιγμή. Η οικονομική αλληλεγγύη σημαίνει για πολλούς ότι η ελίτ του αθλητισμού βοηθάει την βάση του αθλητισμού. Αν δείτε όμως πώς κινούνται οι πόροι, μάλλον κινούνται ανάδρομα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα, τα, κλαμπ, οι λέσχες ε, πληρώνουν για να τροφοδοτήσουν και να υποστηρίξουν τη δράση των ελίτ στον αθλητισμό. Όπως αναφέρεται επίσης, πολλοί πιστεύουν ότι οι ελίτ προωθούν την δράση σε αθλητισμό βάσης, γιατί με τον τρόπο αυτό είναι πιο πολλοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Αλλά δεν υπάρχει καθόλου δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία ότι τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα δημιουργούν περισσότερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη συμμετοχή. Ότι με τον τρόπο αυτό γίνονται περισσότεροι άνθρωποι ενεργοί στον τομέα του αθλητισμού. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο πολύπλοκη από το απλώ να έχουμε μεγαλύτερη ακτινοβολία και ορατότητα των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν στο όραμά μα και σα ζητώ συγγνώμη γιατί έφερα και κάποια τεχνικά βοηθήματα για να σας δείξω τι είναι το όραμά μας. Πέντε αρκουδάκια, τα οποία καταδεικνύουν πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Πέντε μικρά αρκουδάκια, κάθε ένα από τα οποία εκπροσωπεί εκατομμύρια Ευρωπαίους. 40% είναι ενεργοί και 60% δεν είναι τόσο ενεργοί στον αθλητικό τομέα. Και ξέρουν αυτοί που δεν ασκούνται ότι αυτό το οποίο κάνουν είναι επικίνδυνο, ότι η αδράνεια και η, μη, η έλλειψη άσκησης είναι αυτή η οποία οδηγεί σε ασθένειες. Επομένως ο στόχος μας είναι ένα από αυτά τα αρκουδάκια που είναι αδρανές να ανταλλαγεί με ένα αρκουδάκι το οποίο είναι ζωηρό και πεταχτό και θα μας δώσει επομένως άλλους 100 εκατομμύρια που αθλούνται. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήσασταν πολύ καλός παιδαγωγός νομίζω. Αυτά τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιήσατε τα πετύχατε πολύ καλά. Ο κύριος Μισελ Κολούτσι, καθηγητής ε, ε, αθλητικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Τίλμποργκ. First of all, I apologize because I did not bring... Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έφερα αρκουδάκια μαζί μου, αλλά έφερα όμως φοιτητέ αντί για αρκουδάκια. Από όλη την Ευρώπη. On the last row of the In order to speak, him για να μιλάει κανείς και να ονειρεύεται για τις ευρωπαϊκές αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Ποιος μπορεί να κάνει τι. The answers are in the treaty. In the treaty. Ε, και στη συνθήκη πρέπει να διευκρινίζεται αυτό στο 165 και όχι μόνο στο 165. What is the right level of involvement Αλλά για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι στη συνθήκη ο συντονισμός και η υποστήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων τι σημαίνουν άραγε. Σημαίνουν απλά ότι η διακυβέρνηση του αθλητισμού παραμένει πάντα βασική αρμοδιότητα των κρατών μελών από τη μία και των αθλητικών ομοσπονδιών από την άλλη. Βασική ερώτηση είναι το τι, τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν οι εμπλεκόμενοι σε εθνικό επίπεδο και τι μπορούν να ζητήσουν από τα ευρωπαϊκά όργανα και από ποια ευρωπαϊκά όργανα. Ποια Όλοι γνωρίζουμε ότι οι μελέτες που έχουν γίνει ε, διεκδικούν δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, νομική βεβαιότητα, ασφάλεια. Και δεύτερον, αναγνώριση σαν δικηγόρος. Έχω πολλές αμφιβολίες για την ύπαρξη της νομικής βεβαιότητας. Σαν δικηγόρος έχω βασικές αμφιβολίες. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή συντάσσεται ένας κανόνας, ένας νόμος και πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να ερμηνευτεί. Και ποιος θα ερμηνεύσει, ο Μικέλε Κολούτσι, όχι εσείς, όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ερμηνεύσει τον νόμο. Και τι σημαίνει επίσης το να αναγνωρίσουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά. Ο πρώτος ο οποίος έχει ορίσει ένα ειδικό χαρακτηριστικό ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό. Εδώ και χρόνια ήταν ε, στα χέρια μας ήδη από την απόφαση Μπόσμαν. Αλλά ο πρώτος που έδωσε συγκεκριμένους ορισμούς ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, αυτό υπενθυμίζεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης και το Ολυμπιακό κίνημα και οι ομοσπονδίες, οι ελίτ, οι αθλητές κτλ. Και αυτοί δίνουν τους δικούς τους ορισμούς των ειδικών χαρακτηριστικών. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Εγώ έχω ειδικά χαρακτηριστικά, εσείς και εσείς κυρία Πρόεδρε, ειδικά εσείς έχετε ειδικά χαρακτηριστικά. Ποιες είναι οι δυνατότητες τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Δράση. Νομίζω ότι ο Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε μια απάντηση, αλλά Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, δεν συμμερίζομαι αυτή την αίσθηση απογοήτευσης την οποία αναφερθήκατε στην αρχή της ομιλίας σας. Ξέρετε γιατί. Γιατί η συνθήκη βασικά δίνει σε εσά, δίνει σε μας κάτι περισσότερο σχετικά με τις αθλητικές δραστηριότητες. Η συνθήκη αναφέρεται στον αθλητισμό πέραν της οικονομικής διάστασης. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσετε ποτέ το όνομά μου, δεν θα ξεχάσετε ποτέ το πρόσωπό μου. Ποια είναι η εμβέλεια της συνθήκης. Ε, είναι η ειδική συνθήκη για τους επαγγελματίες, είναι η ειδική συνθήκη για τους ερασιτέχνες. Ποιοι είναι οι ερασιτέχνες, είναι αυτοί οι οποίοι ρυθμίζονται από τους κανονισμούς της FIFA, όχι. Ε, ερασιτέχνες είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν για να ευχαριστηθούν οι ίδιοι. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ερασιτέχνες. Εν πάση περιπτώσει τα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα θα πρέπει να αλλάξουν πορεία. και θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στους ερασιτέχνες και όχι μόνο στους επαγγελματίες. Και τώρα να σας κάνω δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Η συνθήκη μας δίνει τη δυνατότητα να συντονίσουμε και να υποστηρίξουμε. Πώς να συντονίσουμε όμως κάτι ή κάποιους Πώς μπορώ να συντονίσω εγώ εσάς αν δεν ξέρω ποιοι είσαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συντονίσει ένα αθλητικό συμβάν μόνο. εφόσον υπάρχει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ή ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο το οποίο πρέπει να έχει τρεις στόχους. Πρώτος στόχος. Δεύτερον, συλλογή πληροφοριών. Ε, σε κάθε ομοσπονδία. Ένας ερασιτέχνης Ιταλός δεν είναι υποχρεωτικά ερασιτέχνης ε, στο Βέλγιο ή στη Γερμανία και οι ορισμοί που δίνει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία στην Ιταλία για το ντόπινγκ ίσως να μην είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο οι αντίστοιχοι ορισμοί και κανόνες της Σουηδικής Ομοσπονδίας συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες, εντοπίζουμε τις αδυναμίες και προσπαθούμε να, να διανύμουμε και να διασπείρουμε σε εισαγωγικά τις βέλτιστες πρακτικές. Να πω επίσης, όχι σαν ακαδημαϊκός, αλλά σαν τον έρασμο. Ήμουν και εγώ κάποτε ε, φοιτητής Εράσμους και ήμουνα υπερήφανος. Ένα από τα πιο σωστά και πετυχημένα προγράμματα της ευρωπαϊκή Ένωσης ήταν το πρόγραμμα Εράσμους. Πάνω από δύο εκατομμύρια φοιτητές πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη για να σπουδάσουν. Γιατί να μην πιστέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο και για τους αθλητές, για αυτούς οι οποίοι είναι ρασιτέχνες αθλητές που το κάνουν για την ευχαρίστησή τους να μπορέσουν να πάνε σε άλλη χώρα να παίξουν. Το ίδιο να γίνει με τους εθελοντές ε, με ένα τέτοιο πρόγραμμα ή για την οργάνωση αθλητικών γεγονότων. Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά, υπάρχουν ήδη στα συμπεράσματα στο Fontainebleau από το 1984. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις βασικές της αξίες θα πρέπει να συμπεριλάβει και τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι βασικό μέσο για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και ευχαριστώ και τους φοιτητές μου που ξύπνησαν χαράματα για να έρθουν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Καλούτσι. Κολούτσι. Εκφράζω την απογοήτευσή μου. Πιστέψτε μου, είμαι 21 χρόνια εδώ πέρα και είμαι ακόμα αισιόδοξη. Έκανα μια, υπέβαλα μια έκθεση στα μέσα της δεκαετίας του 90 με στόχο τότε να μπει ο αθλητισμός συνθήκη. Ε, χρειάστηκε λίγος χρόνος αλλά έγινε. Οπότε δεν απογοητεύομαι, αλλά πρέπει να πω πως απογοητευόμαστε όταν ακούμε ε, το τι μπορούμε να κάνουμε στην πραγματικότητα με το άρθρο για τον αθλητισμό. Ε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα μέσο βεβαίως ε, για να κάνουμε πολλά, αλλά πρέπει να υπάρχει διάθεση. Όχι της Κομισιόν, της Κομισιόν υπάρχει, τους υπόλοιπους στη Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία κτλ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ερωτήσεις βλέπω και σχόλια των βουλευτών. Πρώτα απ' όλα η κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν, προς τον κύριο Πόλγκερ για την πολιτική αντι-doping που είναι νομίζω κομμάτι της ε, ανακοίνωσης Κομισιόν. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία με τον Καναδά για την προστασία των δεδομένων των αθλητών της Ένωσης που πηγαίνουν στον Καναδά χωρίς εγγυήσει ε, για τα δεδομένα αυτά. Δεν υπάρχει ακόμα μια εγγύηση για το ότι δεν πηγαίνουν μετά σε τρίτες χώρες, σε τρίτα μέρη, τα δεδομένα αυτά. Υπάρχει μια ομάδα παρακολούθησης, αλλά βεβαίως το ερώτημα είναι κατά πόσο υπάρχει συνεννόηση με τα κράτη-μέλη και αν υπάρχει κάποια... Εάν κάποιος έλεγχος από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου. Οπότε το ερώτημά μου είναι ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της Κομισιόν στην αναθεώρηση του κώδικα της ε, ΟΑΝΤΑ για αν ε, θα μπορέσουμε εμείς επίσης να έχουμε κάποιο λόγο για τις συζητήσεις μεταξύ Κομισιόν και Γουάντα και τέλος ε, τι σκοπεύει η Κομισιόν να κάνει για την παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου από τον κώδικα της Γουάντα. Ε, καλός αθλητισμός και τα λοιπά, αλλά πρέπει να τηρούνται και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ όλους τους εισηγητές γιατί νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλιά τους και οι παρατηρήσεις τους και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον κύριο όταν ήμουνα πρόεδρος της Ισπανικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία γεννήθηκαν σε μένα κατά τη διάρκεια αυτών των παρουσιάσεων απαντήθηκαν ήδη από μόνα τους. Αλλά υπάρχει και μια νομική αντίφαση μεταξύ αυτού που λέει το άρθρο 165 των συνδικών που μας λέει κυρίως για τον αθλητισμό στη βάση και αυτό είναι οι αθλητικές δραστηριότητες και η υποστήριξή τους που πρέπει να γίνει σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης όταν συζητώ με αθλητικές ενώσεις μου μιλάνε για θέματα που είναι κάπως διαφορετικά. Αυτή θα θέλα να υπάρχει μια καλύτερη μορφή συντονισμού αυτών των δραστηριοτήτων από την πλευρά της Κομισιόν. Γιατί πρόκειται για ζητήματα που για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όταν ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός ο συντονισμός. Για τους μάνατζερ, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν έχουμε εκεί μια απάντηση. Τα στοιχήματα, η ελεύθερη κυκλοφορία των παικτών, η αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων των προπονητών, να υπάρξει κοινή νομοθεσία για μια πλειάδα θεμάτων στην Ευρώπη. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αγώνας κατά της μυσαλλοδοξίας, της διάκρισης, του ντοπαρίσματος. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται από το άρθρο 165, αλλά ενδεχομένως θα προσπαθήσαμε να βρούμε και άλλες νομικές βάσεις και άλλες βάσεις για δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλα άρθρα για να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό. Κάτι ακόμα που είναι επίσης σημαντικό να γίνουν κάποιες χειρονομίες για να δείξουμε ότι η Ευρώπη υποστηρίζει τον αθλητισμό. Παραδείγματος χάρη, η επιτυχία της ομάδος γκολφ της Ευρώπης στο Ryder Cup. Άτομα τα οποία πολλοί ε, πολύ λίγο ασχολούνται με τον αθλητισμό, παρακολουθήσαμε μεγάλο ενθουσιασμό του παίκτε γκολφ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρώπη, οι οποίοι νίκησαν του Αμερικανού. Και έλεγα, γιατί να μην φέρουμε παραγωγή χάρη στο κοινοβούλιο την ομάδα του Ryder Cup με το κύπελο το οποίο κατέκτησαν επαξία. Αυτό μπορεί να δώσει λοιπόν μια μεγαλύτερη ακτινοβολία στην προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τον αθλητισμό. Τέλο, θέλω να πω στην Κομισιόν πρέπει να δείξει θάρρο Ακούω αυτά που λέει η πρόεδρο μα ότι έχουμε κάποια όρια σε επίπεδο νομική βάσης, αλλά θα ήταν χρήσιμο να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα νομικά φράγματα για να μην ε, ματαιωθούν οι προσδοκίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τομέα του αθλητισμού. Ο κύριος Κέλλη. Πρώτα απ' Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Σημαντικό είναι να γίνει σήμερα αυτή η συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής του αθλητισμού. Αλλά κάποιοι είναι κάπως επιφυλακτικοί. Νομίζω πως ο κ. Χίκη είπε πως υπάρχει ο κίνδυνος ε, να έχουμε τελικά το αποτέλεσμα να είναι μόνο μπλα μπλα. Και αν ακούσετε όλα όσα είπε η Κομισιόν για το τι καλύπτει η ανακοίνωση αυτή, τότε υπάρχει ο κίνδυνος ε, να μην καταλήξουμε κάπου. Οπότε σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε σε ορισμένα σημεία και να τα καλύψουμε και να τα καλύψουμε σωστά. Πρώτα απ' όλα ο στόχος ε, των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων που θα δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό μας το 2020 είναι κάτι που μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Θα έχει φοβερά ωφέλη σε όλους τους τομείς της ζωής, από την υγεία, τον αθλητισμό κτλ εάν επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Και θα κολλάει ωραία και με τους στόχους του 2020. Όμως, δεύτερον, νομίζω το να γίνεται σήμερα μια τέτοια συζήτηση όταν γύρω μας έχουμε μεγάλες ε, δυσκολίες να υπογράψουν οι συνάδελφοι τη γραπτή δήλωση για τον αθλητισμό, ε, αυτό είναι ένα άσχημο μήνυμα. Ειδικά όταν μετά την έμφαση που δόθηκε στη συνθήκη Λισαβόνα στο άρθρο 165 και ανέβηκαν οι προσδοκίες, όπως είπε ο κ. Χίκη, και μετά αν εμείς ως βουλευτές δεν υπογράφουμε τη γραπτή δήλωση, αρκετοί τουλάχιστον, τότε και αυτό θα είναι ένα αρνητικό μήνυμα. Ελπίζω λοιπόν στην επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο αρκετοί συνάδελφοι να υπογράψουν. Τέλος να πω πως το Εράσμους για τον αθλητισμό το είχα ε, προτείνει εγώ σε ένα άρθρο πριν από 14 μήνες. Είναι εξαιρετική ιδέα και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Λίγοι στόχοι λοιπόν, να τους επιτύχουμε και να ε, τα κάνουμε σωστά τα πράγματα. Αγαπητοί συνάδελφε, θέλω να τονίσω το θέμα της γραπτής δήλωσης. Δεν έχει σχέση με την Επιτροπή μας. Εγώ είμαι κατά αυτών των γραπτών δηλώσεων. Η δουλειά μας γίνεται εδώ μέσα και σε άλλες συνεδριάσεις ε, ή σε ομάδες, αλλά δεν τις μπορώ αυτές τις γραπτές δηλώσεις. Δεν, δεν θα υπογράψω ποτέ κάτι τέτοιο. Και δεν έχει σχέση, μην αποδίδεται τόση σημασία σε αυτό το πράγμα. Σημασία έχουν τα όσα κάνουμε εδώ πέρα. Ίσως και οι διακομματικές ομάδες. Αλλά για τις γραπτές δηλώσεις, τι να σου πω, είναι χάσιμο χρόνο. Και δεν αφορά εσάς, αφορά τις γραπτές αυτές δηλώσεις. Κυρία Πρόεδρε, ναι, κύριε Κέλλη ορίστε. Υπάρχει μια γραπτή δήλωση Θεωρώ πως αν δεν δημογράψουν αρκετοί συνάδελφοι θα αποστείλουμε το λάθος μήνυμα. Ε, κανείς δεν αναγκάζει κανέναν να το κάνει, αν θέλουν. Ευχαριστώ. Να το ξαναπώ. Δεν είναι το, το μέσο για να κάνουν έτσι οι βουλευτές πολιτικοί. Ας το κάνει, εν πάση περιπτώσει, κανείς αν έχει χρόνο. Εγώ πάντα το ίδιο έλεγα. Λοιπόν, ο, ο αντιπρόεδρος κ. Σουήνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγον ότι τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το θέμα της συνθήκης Λισαβόνας. Εμείς στη Φιλανδία και στις σκανδιναβικές χώρες έχουμε περιορισμένες εξουσίες στους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τον αθλητισμό. Επομένω αυτό περιορίζει και τις δυνατότητες δράσης στον τομέα αυτό και οι πρωτοβουλίε των πολιτών έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ένα πιο σημαντικό ρόλο στι βόρειε χώρε τη Ευρώπη από τι νότιε χώρε τη Ευρώπη, όπου το κράτο ασχολείται πολύ περισσότερο με τα αθλητικά θέματα. Για μας η αθλητική δραστηριότητα και η οργάνωση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ε, εθελοντικές ενώσεις των πολιτών και τους αθλητικούς συλλόγους. Πιστεύω λοιπόν πρέπει να ταινίσουμε με αυτόν τον τρόπο τη αθλητική δραστηριότητα και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη επίσημη ε, αναγνώριση των εθελοντικών αυτών δραστηριοτήτων. Το ερώτημά μου είναι πόσο καλά γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ποικιλία αντιμετωπίσεων που υπάρχουν στα κράτη-μέλη σε σχέση με την αθλητική δραστηριότητα. Αναγνωρίζει και σέβεται αυτήν την ε, πολυπικιλία και με ποιο τρόπο θέλει να προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα σε αυτή την ποικιλία την αθλητική δραστηριότητα. Ευχαριστώ λέει και ο κύριο Τάκουλα. Θα ήθελα και εγώ από τη δική μου πλευρά να υποστηρίξω αυτά που είπε ο προλαλή σα. Αναφέρθηκε το άρθρο 165 από τους ε, ομιλητές του πάνελ. αλλά υπάρχει και μία ασάφεια για, στο άρθρο αυτό για την ιδιαιτερότητα του αθλητικού της αθλητικής δραστηριότητας και πρέπει να διαλευκανθεί αυτό το άρθρο όπως ε, υποσχέθηκε και η Κομισιόν να προχωρήσει σε μία συγκεκριμένη ερμηνεία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι κανόνες πλαισίου που να καλύπτουν την αθλητική δραστηριότητα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να βρούμε μία μορφή καλύτερου ορισμού και μία πολιτική τοποθέτηση για τα θέματα του αθλητισμού ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό που δίνει το Συμβούλιο της Ευρώπης για τον αθλητισμό. Μια δυνατότητα είναι αυτή. Και εμεί θέλουμε να παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τι δραστηριότητέ τη ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα ορισμό ο οποίο θα προσδώσει ασφάλεια δικαίου για τα θέματα αυτά. Επίση, η Κομισιόν δεν έχει ε, ανταποκριθεί στι ε, επιδιώξει για να υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τον αθλητισμό. Οι προετοιμασίες τώρα για το 2012-2013 για αθλητικά προγράμματα ουσιαστικά έχουν ακυρωθεί. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ καλό και οι εκπρόσωποι των αθλητικών ενώσεων και αυτοί δεν θεωρούν ότι καλό να μην χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες που δίδει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και επίσης εγώ ανησυχώ με αυτό που είπατε για την πυραμίδα στον αθλητισμό. Είναι πράγματι αυτό ένα εύστοχο υπόδειγμα. Και θα πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα η ροή κονδυλίων, η ροή πόρων μέσα σε αυτή την πυραμίδα. θα μπορούσε αυτό να είναι ένα υπόδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ισχύει για όλα τα, όλες τις μορφές αθλητισμού. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ πως ειδικά αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπόλγκερ στην αρχή, αρχή για την ανακοίνωση της Κομισιόν μας δείχνει πόσο μεγάλο είναι το εύρος των ζητημάτων που μας απασχολούν στον αθλητισμό το πρόβλημα με το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι αφενός το ότι δεν έχουμε μέσα λεφτά δηλαδή για να εφαρμοστούν όλα αυτά για να επιτύχουμε όλους αυτούς τα σμάσιους στόχους που αναφέρατε σε σχέση με το 2020 και τα λοιπά και αφετέρου ως το είπαμε αυτό και στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες φιλοδοξίες κομισιών στον τομέα της ε, νομοθεσίας, ε, ειδικά όταν είναι να φύγουμε από το άρθρο 165. Υπενθυμίζω εδώ πέρα το αίτημά μας προς την Κομισιόν να ξεκινήσει μια διαδικασία έλεγχου και επιστοποίησης των ε, μάνατζερ των παιχτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε έχουμε μία αντίφαση. Όλους αυτούς τους ωραίους στόχους, αλλά δεν ε, έχουμε τα μέσα για να τους επιτύχουμε. Οπότε το ερώτημά μου προς τους συνδέσμους και τις ομοσπονδίες είναι το εξής. Ο κύριος Χίκη είπε πως δεν είναι αρκετά φιλόδοξη εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το ερώτημα μου είναι ποιες συγκεκριμένες προσδοκίες έχουν οι Ομοσπονδίες από την αθλητική πολιτική της Ένωσης, ειδικά στον τομέα της νομοθεσίας. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Κολούτσι αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του αθλητισμού, ότι δεν μιλάμε δηλαδή για πράγματα που μπορούν να κρυθούν με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Οπότε θα ήθελα κάποια συγκεκριμένα, κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τώρα, για το Εράσμους, όλοι θα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να βρούμε τα κατάλληλα μέσα και θεωρώ πως ειδικά για το μαζικό αθλητισμό πρέπει να το υποστηρίξουμε, όχι στον τομέα των μεγάλων ομάδων Τώρα όσον αφορά το συνθήκη της Λισαβόνας, πράγματι το άρθρο 165 είναι ασαφές, αλλά ακριβώς επειδή είναι ασαφές είναι και μια ευκαιρία και εναπόκειται στην Επιτροπή μας να ορίσουμε το τι θα γίνει με αυτό το άρθρο και πρέπει να συνεχιστεί άρα ε, η σημερινή συζήτηση και να εστιαστούμε σε κάποια θέματα γιατί όπως σας είπα είναι ευρύτατο το φάσμα από τους επαγγελματίες αθλητές, ε, το ντόπινγκ, ε, θα μπορούσαμε εκεί λίγο να εστιαστούμε και να ορίσουμε και να εκμεταλλευτούμε εμείς τα όσα λέει η συνθήκη. Να πούμε πώς εμείς ερμηνεύουμε το άρθρο 165. Ευχαριστώ κύριος Μπόρις από την Πολωνία. Ε, ευχαριστώ, Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους προλαλήσαντες. Είναι γεγονός ότι η πολιτική για τον αθλητισμό δεν έχει καθοριστεί με αρκετή επακρίβεια. Αυτό είναι μια πρόκληση και για μας και για την Επιτροπή μας. Γιατί εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη μιας αθλητικής πολιτικής. Αν υπάρχει όμως το άρθρο 165 στη συνθήκη, αυτό σημαίνει ότι εμεί θα πρέπει να διαμορφώσουμε, να βοηθήσουμε να διαμορφωθεί αυτή η πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Σκολούτσι αναφέρθηκε στην πραγματικότητα τη ε, νομική στην ε, ποικιλία των νομικών ερμηνεών αυτού του άρθρου και έχουν παρουσιαστεί διάφορα υποδείγματα για την αθλητική δραστηριότητα και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Γκαγιά ο οποίος μας παρουσίασε ένα συνολικό υπόδειγμα, ένα ευρωπαϊκό συνολικό μοντέλο για τον αθλητισμό που περιλαμβάνει και τους ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες και τους αθλούμενους βάσεις. Είναι αυτό το υπόδειγμα της πυραμίδας. Αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, υποστηρίξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού βέβαια καθορίσουμε σαφέστερα τι σημαίνει το άρθρο 165. Και αυτά τα οποία ανέφερε και ο κύριο Πόλγκερ δεν ήταν συγκεκριμένοι στόχοι, ήταν περισσότερο ιδέε για το πώ μπορούμε ένα τέτοιο υπόδειγμα να το κάνουμε πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι οι ορισμοί που ανθεσέδωσε ο κύριος Κολούτσι μας δίνουν πολύ καλές οδούς για να συντονίσουμε και να υλοποιήσουμε την πολιτική αθλητισμού στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή είναι η διαδικασία συντονισμού μεταξύ των κρατών μερών πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσθέσει κάτι. Και εδώ είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω στους προδαλήσαντες. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα χώρο για την ευρωπαϊκή πολιτική αθλητισμού με το υπόδειγμα αυτό πυραμίδα το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Αυτό για σας φαίνεται να είναι μια αξιόπιστη οδός. Ευχαριστώ Λεόπλα. Ο Μάρκους Κορέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματι η ακρόαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σε σχέση με το περιεχόμενο και σε σχέση με τη μορφή, την παρουσίαση. Δεν ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα για τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να αναγνωρίσει τον αθλητισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε ότι υπάρχουν διάφοροι τομείς οι οποίοι προκαλούν ενδιαφέρον όπως ε, αυτών που έχουν ε, περιορισμούς κινητικότητας, ε, αθλητισμός και μετανάστες και διάφορα επιμέρους τέτοια στοιχεία. Αλλά Είδαμε επίσης ε, και το θέμα των πόρων που δεν έχουμε και που θα θέλαμε να έχουμε τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό. Να κάνω μία πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε και κάποιος άλλος συνάδελφος, θα ήθελα η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην είναι ένα απλό πλαίσιο το οποίο να απαριθμεί τις δυνατότητες παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε λίγους στόχους, ξεκάθαρους στόχους σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και εφικτούς στην επίτευξή του στόχους. Συνεπώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε τα επόμενα χρόνια να κατευθύνουμε τις αθλητικές δραστηριότητες μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τουλάχιστον σε ένα επίπεδο τις προσδοκίες κάποιων ομοσπονδιών και όχι να μιλάμε για τα πάντα και στην πρακτική να μην κάνουμε τίποτα. Λοιπόν αυτό είναι το αίτημά μου. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να ορίσουμε σωστά συνεπώς τους τομείς παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον γύρω από τον αθλητισμό. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο πρώτος γύρος. Θα ακολουθήσει ο δεύτερο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα δώσω τον λόγο στον κύριο Πόλγκερ. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα οποία ακούστηκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Οι ερωτήσεις ήδη καταδεικνύουν το φάσμα των ζητημάτων που καλύπτει ο αθλητισμός και κείμενεται από ζητήματα χρηματοδότησης μέχρι πολύπλοκα θέματα νομικά και ζητήματα όπως το ντόπινγκ. Θα το τελευταίο γιατί ήταν το πρώτο ερώτημα το οποίο τέθη από την κυρία Μποσκούρτ για το ντόπινγκ. Είναι σαφές πως το άρθρο 165 μας δίνει ένα μοχλό για να δράσουμε για το ντόπινγκ. Γιατί μιλάει ρητά για την σωματική και ηθική ακαιρεότητα των αθλητών. Ξεκάθαρη αναφορά στο ντόπινγκ. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Το ντόπινγκ ρυθμίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο από την Γουάντα που βρίσκεται στο Μοντρεάλ, στον Καναδά. αποτελείται από εκπροσώπους του αθλητισμού και των κυβερνήσεων. 50-50. Η Ευρώπη έχει πέντε έδρες στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. Δύο είναι για το Συμβούλιο της Ευρώπης και τρεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει επίσης μια εκτελεστική επιτροπή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μέλος. Μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω, πριν τη θέση ενισχύ της Λισαβόνας, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπόταν από τρεις υπουργούς, από τον υπουργό της χώρας που έχει την Προεδρία. Ένα από τα προβλήματα του συστήματος το επεσήμανε η κυρία Μποσκούρτ. Δηλαδή δεν υπάρχει συνέχεια. Όταν υπάρχει συνεχής εναλλαγή σε ένα θέμα στο οποίο χρειάζονται δίκτυα, γνώση, επιρροή, ε, η Ευρώπη καθίσατε αδύναμη. Στο συμβούλιο αυτό του Ιδρύματος. Επιπλέον, τα μέλη πηγαίνουν εκεί χωρίς καμιά εντολή. Δεν υπάρχει μηχανισμός για να τους δοθεί κάποια εντολή. Σε πολλούς άλλους τομείς, όταν εκπροσωπούν οι Υπουργοί την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εντολή από το Συμβούλιο. Και τώρα πρέπει με τη Λισαβόνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνενέσει, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει εντολή. Οπότε μιλάνε σε προσωπικό επίπεδο, δεν εκπροσωπούν την Ένωση. Οπότε η Ευρώπη στη Γουάντα είναι σε ε, άσχημη θέση. Ανεξάρτητος του ότι πληρώνει σχεδόν το μισό προϋπολογισμό της, της δεν έχει το 50% της ε, επιρροής που θα έπρεπε να έχει. Έχουμε λοιπόν, όπως είπα, εκπροσώπους της Βελγικής Προεδρίας. Η Βελγική Προεδρία το είδε αυτό το πρόβλημα. Προσπάθησε να δώσει μια λύση. Υπάρχει μια συνεδρίαση του Συμβουλίου αυτού την ε, ερχόμενη εβδομάδα και προσπάθησε να το συντονίσει αυτό η Κομισιόν καθώς αυτό είναι υποχρέωση από συνθήκη. Πρέπει να συντονίζονται σε διεθνή βήματα τα κράτη-μέλη και σε σχέση με το δεδομένο, το, με το κοινοτικό κεκτημένο το οποίο αφορά παραδείγματος χάρη όπως αναφέρθηκε την προστασία των δεδομένων. Βεβαίως ο Καναδάς είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τα δεδομένα αυτά μπορούν να πάνε ε, οπουδήποτε στον κόσμο και βεβαίω αυτό αντιβαίνει και το γράμμα και, το... και στο πνεύμα της ε, Ευρωπαϊκής Οδηγίας για δεδομένα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα με τον κώδικα της Γουάντα αλλά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μέχρι να υπάρχει κάποιο μέσο για τον συντονισμό. Η Βελγική Προεδρία όσον αφορά τον συντονισμό έκανε ένα βήμα γιατί απόψε η Υπουργοί Αθλητισμού θα υιοθετήσουν συμπεράσματα του Συμβουλίου για αυτό το οποίο λέγαμε συντονισμό της Ένωσης πριν τις συνεδριάσεις ε, του Συμβουλίου του Ιδρύματος της Οάντα. Αντιλαμβάνομαι επίση πω η Ουγγρική και η Πολωνική Προεδρία είναι έτοιμε να δουν το ζήτημα τη εκπροσώπηση. Γιατί τώρα που ο αθλητισμό αναφέρεται επισήμω στη συνθήκη, το Συμβούλιο μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα όπου θα έχουμε πραγματικά αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους. Αυτά για το πρώτο. Προφανώ δεν θα με απασχολήσουν τόσο πολύ όλα τα ζητήματα. όλε οι ερωτήσεις. Να αναφερθώ στο τι δυνατότητες μας δίνει το άρθρο 165 γιατί νομίζω πως θα ορίσει και τις φιλοδοξίες θα έχουμε. Το άρθρο 165 η διάταξη για τον αθλητισμό είναι σε ένα άρθρο περί εκπαίδευση, όπως ξέρετε. Το συγκεκριμένο αυτό άρθρο μας δίνει δύο μέσα για να κάνουμε κάποια πράγματα. Το ένα είναι οι συστάσει του Συμβουλίου, αλλά είναι συστάσεις με βάση μια πρόταση της Κομισιόν. Και Το κοινοβούλιο δεν έχει κανένα ρόλο εκεί πέρα και αυτό είναι μια δυναμία τη συνθήκη εδώ πέρα. Αντικατοπτρίζει βεβαίως ε, τις απόψεις των συντακτών της συνθήκης ότι αυτά τα θέματα είναι θέματα επικουρικότητας. Άρα το αποτέλεσμα είναι πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει και αυτό είναι κρίμα. Γιατί οι συστάσεις μπορούν να διαμορφώσουν την εφαρμογή των κανόνων. Μπορούν δώσουν κατευθυντήριες γραμμές ε, και στους δικαστές ε, και στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή. Δυστυχώς η οδηγία δεν προβλέπει συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Τι άλλο ε, περιέχει το 165. Μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε προγράμματα. Και εδώ πέρα βέβαιω έχει πλήρη ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είμαστε στη συναπόφαση. Συναποφασίζει τα προγράμματα το Κοινοβούλιο δυστυχώς η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετέθην ισχύ σε μια πολύ ακατάλληλη στιγμή από πλευράς οικονομικής. Το άρθρο 165 μας δίνει μια νομική βάση αλλά όχι προϋπολογισμό. Αρχικά η Κομισιόν θεωρούσε πως θα ήταν καλή ιδέα να έχουμε ένα μίνι πρόγραμμα για να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ 2014 και των ε, προπαρασκευαστικών δράσεων ε, που ψήφισε η Επιτροπή σας μέχρι το 2011, αλλά ανακαλύψαμε πως στον τίτλο του προπολογισμού εντό του οποίου κινούμαστε δεν υπάρχει πλέον περιθώριο. Δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή. Τα λεφτά πρέπει να τα πάρουμε από κάπου αλλού. Από το Εράσμους ας πούμε. Δεν νομίζω να σας άρεσε αυτό. Θα θυμάστε. Κυρία Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε, ένα από τα τελευταία πράγματα που κάναμε μαζί όταν ήμουν υπεύθυνο για τα ΜΜΕ ήταν το πρόγραμμα Media Mundus που πέρασε από τη συναπόφαση σε χρόνο ρεκόρ γιατί δεν υπήρχε χρόνος. Τελείωναν τα λεφτά και μιλούσαμε για 3 επί 5, 3 φορές 5 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα βρούμε λοιπόν τα, τα λεφτά εδώ πέρα. Ακόμα λοιπόν και με τα προγράμματα τα οποία είναι πλήρως αναπτυγμένα ε, δεν θα μπορέσουμε ήδη από του χρόνου, από την αρχή τουλάχιστον, να τα εφαρμόσουμε. Γιατί οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 11 ξέρετε ότι κατέρευσαν προχθές. Δεν έχουμε προϋπολογισμό για το 11 και εσείς σαν βουλευτές γνωρίζετε τα δημοσιονομικά προβλήματα αυτό το οποίο συνέβη για το 2011 είναι θα έλεγα πρελούδιο στο τι αναμένεται για τις συζητήσεις για, τις, ε, για, το πολιετές πλαίσιο προγραμματισμού μετά το 2014. Θα δοθεί μια πολύ σκληρή μάχη για τις δημοσιονομικές προοπτικές και θα υπάρξουν πιέσεις για να απαλλαγούμε από το Εράσμους, από πολιτιστικά προγράμματα, από προγράμματα μέσων ενημέρωσης όπως το Μέντια. Θα υπάρξουν πιέσεις για νέα προγράμματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει ε, κάποιες μελέτες ε, προοπτικές για τις επιπτώσεις που θα έχουν ε, τα προγράμματα για τον αθλητισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πεπισμένη για τη χρησιμότητά του η κυρία Βασιλείου και θα θέλαμε βέβαια να κρατήσουμε τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο τον κοινοτικό προϋπολογισμό αν και κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο θα είναι δύσκολο κάποιο νέο πρόγραμμα να γίνει δεκτό αν και πιστεύουμε πλήρως στην αξία ενός προγράμματος στήριξης του αθλητισμού. αυτά σε επίπεδο κινήτρων. Τι να πω τώρα για κάτι που αναφέρθηκαν κάποια μέλη σας γύρω από τα υπόλοιπα άρθρα. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε τον αθλητισμό και σε άλλους τομείς στα πλαίσια του λεγόμενου mainstream όπως ε, η εκπαίδευση, η νεότητα, σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα ο αθλητισμός στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος δράσης για τη νεότητα, το 11 και το 12. ο υπεύθυνο Επίτροπος για τα διαφορετικά ταμεία και θα φαίνεται αυτό στην ανακοίνωση της Επιτροπής είναι δεκτικός για τη χρηματοδότηση αθλητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια των διαφορετικών ταμείων. Αλλά κάποιες νομικές ρυθμίσεις στη συνθήκη, σε σχέση με τη συνθήκη, είναι αντιδραστικά σε εισαγωγικά, δηλαδή ενεργοποιούνται από αυτούς οι οποίοι ε, προσφεύγουν στο δικαστήριο εναντίον των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δημιουργούνται συγκεκριμένα θέματα. Όπως είπε και ο καθηγητής Κολούτσι, τι θα πει ειδικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει εμείς να τα ορίσουμε. Οι λήπτες αποφάσεων μέσω της διαμόρφωσης της πολιτικής στην οποία προχωρούν μπορούν να επηρεάσουν την ερμηνεία όρων όπως τα ειδικά χαρακτηριστικά. Έχει υπάρξει μια περίπτωση στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η περίπτωση Ολιβιέ Μπερνάρ, μια περίπτωση ποδοσφαιρικής μεταγραφής και εκεί το δικαστήριο έκανε ό,τι μπορούσε για να αναφερθεί στον όρο ειδικά χαρακτηριστικά. Δεν ήταν υποχρεωμένο να το κάνει, αλλά επέλεξε να το κάνει. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό μήνυμα το δικαστήριο για το μέλλον. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτό, ειδικά χαρακτηριστικά, για να μπορέσουμε να θεμελιώσουμε θα έλεγα μια σταθερή νομική ερμηνεία και του πρωτογενού δικαίου και των οδηγιών και της νομολογίας ειδικότερα. Αν θέλει κάποιος από τους εμπειρογνώμους να κάνει κάποια σύντομη παρατήρηση, κάποιο σχόλιο ή αν θέλει να προσθέσει κάτι μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Αλλιώς θα συνεχίσουμε με τους συναδέλφους αν θέλουν να θέσουν ερωτήματα. Σύντομα όμως, ε μην ανησυχείτε, δεν θέλω να με ξανακτυπήσετε με το σφυρί σας. Ένα από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα είναι ότι είμαστε η μόνη ήπειρος που δεν έχουμε ε, αγώνες υπηρωτικούς ολυμπιακού χαρακτήρες όπως υπάρχουν, χαρακτήρα όπως υπάρχουν στην Ασία και στην Αφρική. Έχουμε αγώνες για τους νέους βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή ε, δεν μας δείχνει αυτό γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν πανευρωπαϊκοί αγώνες ολυμπιακού χαρακτήρες. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει κάτι τέτοιο. Είναι εξελίξει, συζητήσει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Οι υπηρετικοί Ολυμπιακοί αγώνε λοιπόν στην ε, Ευρώπη θα μπορούσαν να συνδυαστούν θαυμάσια με αυτά που θέλει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ, λέγει Πρόεδρο. Και τώρα, από τη Σλοβανία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήθελα να αντιμετωπίσω τα ερωτήματα αυτά για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ως Ευρώπη τα θέματα του ντοπαρίσματος και να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρώπης στην Επιτροπή της ΟΑΝΤΑ. Η απάντηση έχει δοθεί εν μέρη ήδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αν είχε ένα εκπρόσωπο ένα μόνιμο εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ένα εκπρόσωπο του Συμβουλίου και της Κομισιόν, αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό για να ενισχυθεί η εργασία μας στον τομέα αυτό. Εγώ ήμουνα ε, μέλος της Οάντα ως ε, εμπλεκόμενος στον αθλητισμό και βλέπω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ε, παρουσία εκεί. Η επιρροή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ περιορισμένη στη Γουάντα σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου όπως παραδείγματος χάρη η Αυστραλία. Και εδώ θέλω να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχουν έρευνες για το πάρισμα ή μάλλον οι έρευνες για το ντοπάρισμα είναι συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα των αθλητών και οι κυρώσει οι οποίε επιβάλλονται επίση. Ένα ακόμα ερώτημα για τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή, τον κύριο Χίκη. Από ποια χρονική στιγμή θα έχουμε και τη δυνατότητα οι ενώσεις σκακιστών να συμμετέχουν. Κύριε Μακάκ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους που πήρατε το λόγο σήμερα όλους τους εμπειρογνώμονες και από τις Ολυμπιακές Επιτροπές και από την UEFA και ευχαριστώ και τον κύριο Κέρκη και τον κύριο Κολούτσι που αναφέρθηκαν και στον τεχνικό αθλητισμό. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει σε σχέση με τον τεχνικό αθλητισμό, τον λαϊκό αθλητισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ερωτήσει μου είναι περισσότερο στραμμένε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα θέματα της χρηματοδότηση. Έχουμε αυξήσει τι προσδοκίε με τη συμπερίληψη του αθλητισμού στη συνθήκη και υπάρχουν ορισμένα κενά εδώ τα, στα οποία αναφερθήκατε. Όχι μόνο δεν υπάρχουν εγγυήσει για τη μελλοντική χρηματοδότηση, αλλά υπάρχουν και προοπτικές απόσυρσης από τη χρηματοδότηση αθλητικών προγραμμάτων, αν και λέτε ότι εκεί υπάρχουν κάποιες προσπάθειες αποκατάστασης των προσπαθειών αυτών. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες εγγυήσει για αυτή την προσπάθεια και πότε θα έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Σχετικά τώρα με την εμπλοκή ε, των ενδιαφερομένων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρώσει κανείς ε, σε αυτές τις συζητήσεις όλα τα αθλήματα. Πώς εσείς μεθοδεύετε τις διαδικασίες αυτές διαβούλευσης. Νομίζω ότι ακόμα και τα λεγόμενα μειονοτικά αθλήματα δεν έχουν την δυνατότητα να ακούγονται οι ιδέες τους σχετικά με το τι μπορούν να προσφέρουν στην, στο σύνολο της δραστηριότητας. Ευχαριστώ. Κώστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξετίμησα δεόντως τις ομιλίες των εμπειρογνωμόνων σήμερα το πρωί, ήταν πολύ πλούσια. Τρεις ερωτήσεις σχετικά με το 165. Αφήνει πολλές εκκρεμότητες και περισσότερες θα έλεγα ερωτήσεις από όσες απαντήσεις. Ας πούμε ότι το άρθρο αυτό δίνει την δυνατότητα και νομιμοποιεί τις ευρωπαϊκές αρχές να θεωρήσουν ότι ο αθλητισμός μπορεί κάλλιστα να είναι τμήμα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Σημασία μεγάλη έχει αυτό. Δεν υπάρχει επίσης ε, ε, αμφιβολία ότι υπάρχει μια οριζόντια διάσταση στον αθλητισμό, κάτι το οποίο θα έλεγα μπορεί να είναι χρήσιμο σε επίπεδο εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας κτλ. Σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά. Και εμείς και η Επιτροπή και οι αθλητικές οργανώσεις πρέπει μετά τη Λευκή Βίβλο να βρούμε πού μπορούμε να εντοπίσουμε αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους. Υπάρχουν δικαιώματα, ξέρετε τώρα, τα οποία είναι εμπεριστατωμένα, θα έλεγα, και τεκμηριωμένα μέσα στη συνθήκη της Ρώμης, όπως το δικαίωμα στην υγεία. Και εδώ θα πρέπει, σε αυτό το πλαίσιο, να διασφαλίσουμε την κινητικότητα στον αθλητισμό, ξεπερνώντας την αρχή της επικουρικότητας και επιδιώκοντας μια καλύτερη εναρμόνιση των πλαισίων αυτών στο εσωτερικό της Ένωσης. Το θέμα των πόρων είναι βέβαια καθοριστικό, αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με τον Επίτροπο για τις Περιφερειακές Πολιτικές έτσι ώστε ήδη από το 2011 να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες πολιτικές όπως ε, που στοχεύουν στην αύξηση της αθλητικής δραστηριότητας, πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να είναι μετρήσιμες και οι οποίες θα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα μέσω των διαφορετικών ταμείων. Και όχι μόνο από δημόσιους οργανισμούς αλλά και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες κάτι που μπορεί να, σας, ε, να το θεωρήσετε αστείο, αλλά υπάρχει ένας προϋπολογισμός που διαμορφώνονται σε αιτήσια βάση από τα λαχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στην Ιταλία το κάνουμε αυτό και παίρνουμε λεφτά από τα λαχεία για τα πολιτιστικά αγαθά να πηγαίνει και στα αθλητικά λεγόμενα σε εισαγωγικά. Λοιπόν, σχετικά με τη γνωμοδότηση φύσας. Πράγματι η ιδέα των Ολυμπιακών Ευρωπαϊκών Αγώνων μου αρέσει. Η ιδέα επίσης της αθλητικής πρωτεύουσα είναι και αυτή μια καλή ιδέα. Νομίζω ότι αυτό το πρότυπο διακυβέρνησης, το οποίο αντιμετωπίζεται από άλλους με κριτική, από άλλους ιδιαίτερα θετικά, προκαλεί συζητήσεις, μεν, αλλά είναι κάτι που ενδιαφέρει τις τοπικές αρχές γιατί η governance όπως λέμε δεν μπορεί να είναι μόνο οριζόντια αλλά αφορά γενικά όλα τα επίπεδα της πυραμίδας. Οι πόλεις, οι τοπικές αρχές που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό είναι σε θέση νομίζω να χρησιμοποιήσουν και τα διαφορετικά ταμεία για να επιτύχουν το στόχο τους. Τσένι σύνα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού οι οποίοι μα έκαναν παρουσιάσει από το πάνελ. Καταλαβαίνω την ανησυχία η οποία διατρέχει αυτή τη στιγμή τον κόσμο του αθλητισμού σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των μεροντικών αθλητικών δραστηριοτήτων και είναι ελπίδα μου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει το καθήκον της και θα μπορέσει να μας παρουσιάσει εν καιρό ένα πλήρες πρόγραμμα. Γνωρίζω ότι ο προϋπολογισμός μας είναι περιορισμένος, όπως είναι και ο προπολογισμό των κρατών μελών για τα θέματα τα αθλητικά. Αλλά θα έχουμε πάντα αυτά τα προβλήματα και μέσα σε αυτά θα πρέπει να αναπτύξουμε κάποιες δραστήσεις. Υπάρχει πρόβλημα με τη μετάφραση από τα πολωνικά. Επομένως, πρέπει κάτω από τέτοιες ε, συνθήκες να συνεχίσουμε. Υπάρχει πρόβλημα στα γερμανικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά, λέει η πρόεδρος. Παρακαλώ. Δεν θέλουμε λοιπόν να, δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουν καλύτεροι καιροί, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να δράξουμε τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το ερώτημά μου προς την Κομισιόν τώρα είναι το εξής. Τι ακριβώς θέλει να... Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος, δυστυχώς. Μα υπάρχει μετάφραση από τα... προς τα γερμανικά αυτή τη στιγμή. Ίσως μόνο στην πρώτη σειρά υπάρχουν προβλήματα. Μπορείτε να μεταφερθείτε ίσως σε κάποια άλλα έδρα, αν θέλετε. Η ελπίδα μου λοιπόν, όπως έλεγα προηγουμένως, ήταν ότι... ότι θα μπορέσει να ε, αποκατασταθεί η διερμηνία και στην πρώτη σειρά. Τι θέλει να κάνει λοιπόν η πρώτη η, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει με προγράμματα όπως είναι η νεότη σε δράση, με τα προγράμματα πλαισίου για την έρευνα, για τα διαφορετικά ταμεία, για το πρόγραμμα Δάφνη, να κάνει προσπάθειες για να υπάρξει καλύτερη υποστήριξη του αθλητισμού στην Ευρώπη. γιατί ο αθλητισμός παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Μαθαίνει τους ανθρώπους ο αθλητισμός να μην σκέφτονται με τρόπους αποκλειστικούς και να μην περιθωριοποιούν κοινωνικές ομάδες, προωθεί την ε, ε υγεία και την ε, ανταγωνιστικότητα λοιπόν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε ο αθλητισμός. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι εσείς κυρία Πρόεδρε εκφραστήκατε τόσο αρνητικά για την ε, δήλωση 62, τη γραπτή δήλωση 62, η οποία έχει να κάνει με την υποστήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, του μαζικού αθλητισμού. Είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλους τους αθλητικούς φορείς. Ε, θέσε το ερώτημα ο κ. Κολούτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε για τον εραστεχνικό αθλητισμό. Εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις εραστεχνικές ενώσεις με τη δράση της ε, Επιτροπής μας και των διαπαραταξιακών ομάδων, αλλά και με την υπογραφή της γραπτούς δήλωσης 62. Και ελπίζω ότι και η πρόεδρος θα κατανοήσει την ανάγκη να υποστηριχθεί ε, αυτή η γραπτή δήλωση όπως έχουν υποστηρίξει αυτή τη δήλωση ήδη 125 συνάδελφοι. Θα ήταν λοιπόν πολύ θετικό να συνταχθεί μαζί μας και η κυρία Πρόεδρος και να υπογράψει αυτό το ψήφισμα γιατί είναι δικό μας αυτή τη γραπτή δήλωση γιατί προέρχεται από εμά. Κοιτάξτε, ε, δεν έχει αυτή η δήλωση, δεν έχει καμία σχέση με την ουσία. Μπορεί να είναι εργασιοθεραπεία, αλλά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό δεν τα υπογράφω αυτά. Αν θέλετε εσείς, συνεχίστε. Ευχαριστώ. Ε, εκεί πέρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φύγαν όλοι. Ε, κύριος Μπάγκο. ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους δύο οργανωτές ε, για την ακρόαση αυτή. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ε, σε τρία πράγματα θα ήθελα να φερθώ. Πρώτα απ' όλα ακούστηκε πως 60% από τα 400 εκατομμύρια δεν κάνουν κανένα άθλημα και πρέπει να κινητοποιήσουμε 100 εκατομμύρια πολίτες. Το ερώτημα μου είναι ποιος μπορεί να κάνει τίποτα εδώ πέρα στον τομέα αυτόν. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα μια πρόταση γι' αυτό. Ε, μια ερώτηση στην Ουγγαρία, παραδείγματο χάρη, έχουμε μια βάση δεδομένων στο διαδίκτυο από το Υπουργείο Αθλητισμού και μπορεί κάποιος να κάνει θεματική αναζήτηση ποιοι σύλλογοι υπάρχουν, ποια γήπεδα, ποιες εκδηλώσεις και ε, αυτό μπορεί να γίνει έτσι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν υπάρχει η πρόθεση. Γιατί το θέμα είναι το πώς και δεν ξέρουμε βέβαια πώς αυτό είναι το θέμα το πώς θα κάνει κανείς αθλητισμό Εξάλλου, όπως ξέρετε, σε 40 μέρες θα έχουμε Ουγγρική Προεδρία και είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε αυτά τα ζητήματα. Είμαστε υπερήφανοι στην Ουγγαρία για το ότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές ε, χώρες ε, στην Ευρώπη με πρόεδρο Ολυμπιονίκη και ο Υπουργός Αθλητισμού είναι στην δική μας ε, κοινοβουλευτική ομάδα επίσης, οπότε νομίζω πως θα έχουν πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τρίτο ερώτημα, συμπλήρωση. Αναφέρθηκε η δυνατότητα ενός εράσμους για τον αθλητισμό και η Κομισιόν εδώ πέρα έχει ε, κινητοποιηθεί και αρχές Απριλίου υπάρχει ένα συνέδριο στη Βουδαπέστη ίσως να μην το ξέρουν ακόμα τα μέλη της Επιτροπής αλλά νομίζω πως θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο γι' αυτό θέλουμε να αποκτήσει σημαντικό ρόλο ο αθλητισμός στο Εράσμος. Ευχαριστώ Μπέλετ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσουμε την κοινή μας δυσφορία και απογοήτευση γιατί δεν θα έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα του χρόνου γιατί δεν έχουμε προϋπολογισμό. Αυτό δεν είναι εναντίον αυτής της Βελγικής Προεδρίας που λέγω, αλλά εναντίον των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα ε, των αθλητικών, των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό στην Ευρώπη. Ας συγκεντρώσω τώρα την προσοχή μου στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ε, άμεσο μέλλον. Καταρχάς, ε, οικονομική σταθερότητα των ομάδων και των εραστεχνικών και κυρίως των επαγγελματικών. Πολλές από τις ομάδες αυτές, από τους συλλόγους αυτούς, αντιμετωπίζουν υπαρξιακά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται και σε επίπεδο UEFA αλλά και σε επίπεδο άλλων αθλητικών οργανώσεων ε, σχετικά με την αδειοδότηση των συλλόγων. Νομίζω ότι αυτό είναι προϋπόθεση για το σωστό ανταγωνιστικό fair play στον αθλητισμό. Πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα και στις χαμηλές κατηγορίες και στις υψηλές σχετικά με το ίδιο θέμα νομίζω Πρόεδρε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση της εκπαίδευσης των τοπικών θα έλεγα δραστηριοποιούμενων στον αθλητισμό. Κάποτε όλα αυτά ρυθμίζονται σε τοπικό επίπεδο, τώρα μέσω της UEFA και των άλλων ομοσπονδιών υπάρχει μια γενικότερη ρύθμιση των κανόνων των αθλητικών δραστηριοτήτων. Πρέπει λοιπόν οι ομάδες να τους δοθούν κίνητρα, να χρησιμοποιήσουν σωστά τα νομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και το 165 εδώ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο και γενικότερα για την παιδεία και την αθλητική παιδεία και δίνει την δυνατότητα στις ομάδες να επενδύουν αρκετά τα τοπικά νιάτα τους, στις τοπικές πηγές θα έλεγα έβρεσης παικτών αλλά ταυτόχρονα να υποστηρίζονται οι ίδιοι αυτοί σύλλογοι οικονομικά από τις οργανώσεις, τις ομοσπονδίες κτλ. Κυρία Τρίπελ, αγαπητοί συνάδελφοι, ω μέλο της ομάδα διαπραγματεύση για τον προϋπολογισμό του 2011 και επέκεινα, ήθελα να σας πω ότι δεν είναι σαφές τι θα προκύψει τώρα στα θέματα του προπολογισμού ίσως θα ακολουθεί μια ταχεία διαδικασία. Αν δεχθεί να αλλάξει άποψη το Συμβούλιο, μπορούμε να έχουμε ένα προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους. Δεν έχει αποφασιστεί τίποτα μέχρι τώρα. Αλλιώς θα έχουμε τα προσωρινά δεκατημόρια τουλάχιστον στην αρχή του 2011 και ελπίζουμε ότι αργότερα, το Μάρτιο ή αργότερα, θα έχουμε ένα νέο προϋπολογισμό για το 2011. Όλα εξαρτώνται από τη στάση που θα κρατήσει το Συμβούλιο και πρέπει να κατανοήσετε γιατί το Κοινοβούλιο και η ομάδα διαπραγματεύσεώς μας ήταν τόσο στεναρή στη στάση της. Γιατί όλα αυτά που έχουμε συζητήσει για τον αθλητισμό είναι τμήματα των νέων αρμοδιοτήτων που μας έδωσε η συνθήκη της Λισαβόνας. Η πολιτική μάχη με το Συμβούλιο είναι για το αν θα πάρει το Συμβούλιο στα σοβαρά της συνθήκης της Λισαβόνας ή όχι. Κάποια κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμοι να το πράξουν αυτό. Δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις νέες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου σοβαρά κάτω χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα και εμεί ω ομάδα διαπραγμάτευση και συνδιαλλαγή για τον προπολογισμό έχουμε δεσμευτεί να διασαφηνίσουμε ότι δεν είναι μονάχα θέμα θεσμική ισορροπία, αλλά πρόκειται για τον μελλοντικό πολιτικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του απαραίτητου πόρου για να καλύψει αυτά τα νέα καθήκοντα σε επίπεδο πληρωμών ο προϋπολογισμός τη Ευρωπαϊκής Ένωση είναι κάπου 130 δισεκατομμύρια. Εάν τον διατηρήσουμε σε αυτό το επίπεδο θα είναι ήδη επιτυχία γιατί ο κ. Κάμερον από το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη ανέφερε να μειώσει κατά 0,8% τον προϋπολογισμό, δηλαδή να χάσουμε σχεδόν 13 δισεκατομμύρια Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να περικοπούν και να ψαλιδιστούν πολλά προγράμματα, πολλές πολιτικές και καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα έχουμε στον τομέα της, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, ακόμα και στα διαφορετικά ταμεία και στη γεωργία θα έχουμε προβλήματα, κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η πολιτική απόλυξη ενός τέτοιου εγχειρήματος. Ξέρω ότι το UKIP και πολλά άλλα κόμματα υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα μια μάχη για τις πολιτικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στους κόλπους του Συμβουλίου μεταξύ 100 μερών και σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Αυτά ήθελα λοιπόν να τονίσω και να πω επίσης ότι αυτά που είπε ο Μικέλε Καλούτσι είναι πάρα πολύ σημαντικά για Να μπορέσουμε να δώσουμε σάρκα και γνωστά στο άρθρο 165, να κάνουμε σαφέ ότι είναι ένα άρθρο το οποίο καλύπτει τα θέματα του συντονισμού μεταξύ χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μου αρέσει και αυτή η ιδέα του έρασμου για τον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμό έχει και οικονομική επίπτωση, αλλά πάρα πολλοί θέλουν να ξεπεράσουν απλώ το θέμα τη οικονομική επιτυχία και να εμπλέξουν περισσότερου ανθρώπου, να κινητοποιήσουν περισσότερο του ερασιτέχνες Επομένως και από πολιτική έποψη, αν είμαστε έτοιμοι και ικανοί να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και την αναψυχή και την ε, αθλητική εραστικνική δραστηριότητα, αυτό δεν είναι πολύ θετικό. Αυτά από την κυρία Τρίπλ και τώρα. Ευχαριστώ μας για τον προπολογισμό. Ευχαριστώ συντονιστή ε, του προπολογισμού εδώ στην Επιτροπή αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Πόλκερ είναι κάτι το οποίο θεωρώ πως πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αν κατάλαβα καλά, είχαμε ένα έλλειμμα εδώ πέρα, θέλαμε 10 εκατομμύρια, πήραμε 3 και αν ε, είναι έτσι η κατάσταση έχουμε κάποιο περιθώριο έλιγμων δεν είναι πως έχουμε παραμεριστεί και ξεχαστεί τελείως. Χρειάζεται λοιπόν κάποια πολιτική βούληση. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση, αλλά δεν είναι πως δεν έχουμε και καμία επιλογή, απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Θα είμαι σύντομος. Ε, δεν ε, είμαι ειδικό ε, στα του αθλητισμού, αλλά είμαι ένας πολίτης. Και ως πολίτης συμφωνώ πλήρως με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κολούτσι. Θεωρώ πως η πολιτική μας, το μαζικό αθλητισμό θα είναι ναι, να έχει ένα προληπτικό ρόλο. Όσον αφορά δε, τον επαγγελματικό αθλητισμό, εκεί πέρα μιλάμε για επιχειρήσεις. Και εκεί πέρα δεν χρειάζεται να παίξουμε τέτοιο ρόλο στο επαγγελματικό αθλητισμό. Δεύτερον, Ε, στην αίθουσα σήμερα ε, βρίσκεται ο κ. Βιλεμπέικοφ, ο Βούλγαρος υπουργό Αθλητισμού. Και θα σήμουν ευγνώμων, εάν του επιτρέπατε, να μας πει και αυτός τις απόψεις του. Ευχαριστώ. Okay. Thank you very much, but we have experts and we have the commission. Ευχαριστώ. Έχουμε εμπειρογνώμονε, έχουμε την Κομισιόν, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο όμω. Θέλω να χαιρετήσω λοιπόν την παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού τη Βουλγαρία. Σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα και για το γεγονό ότι παρακολουθείτε όλα αυτά τα οποία λέμε. Θα, παρακαλώ, θα σα παρακαλούσα να τα χρησιμοποιήσετε και το απόγευμα που θα συναντηθείτε στο Συμβούλιο των Υπουργών με του ομολόγου σα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια, υπάρχουν κάποια αντιφατικά στοιχεία, αντιφατικές πληροφορίες για τον προπολογισμό. Ορισμένοι το αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό με, μέσα σε ένα ζωφερό κλίμα, άλλοι θεωρούν ότι αυτό είναι μια ευκαιρία. Βέβαια, έχουμε μεγάλες δυσκολίες γι' αυτό. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε να κάνουμε εμείς σαν Επιτροπή πρέπει να είναι σαφές όλα αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέροντα, ήταν συναρπαστικά. Υπήρξαν πολλαπλές απόψεις για τα θέματα αυτά, αλλά για μένα, εάν θέλουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές από το 2014 και μετά, πρέπει να είμαστε σαφείς μέσα στην Επιτροπή μας για το ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και τι θέλουμε να διεκδικήσουμε. Και νομίζω ότι έχουμε δύο ουσιαστικά παρατάξεις αν, όπως είπε ο κ. Μπέλετ, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στον επαγγελματικό αθλητισμό, επομένως και την νομοθεσία για τον ντόπινγκ, ή αν, από την άλλη μεριά, θέλουμε να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την αθλητική δραστηριότητα σε επίπεδο βάση, σε επίπεδο τοπικό και να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες σε επίπεδο βάση και εραστεχνικό, που είναι και δική μου προτεραιότητα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και θα προσποριστούμε σημαντικά πλεονεκτήματα από τέτοιες δραστηριότητες και στον τομέα της κοινωνικής συνοχής το να έχονται όλοι μαζί και νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορεί να προκύψει από όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα είναι ότι θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε ως Επιτροπή μια περαιτέρω συζήτηση για το ποιες είναι οι προτεραιότητες ώστε όταν χρειάζεται να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα έχουμε καμία ευκαιρία ε, καμία ευκαιρία να πάρουμε χρηματοδότηση για οτιδήποτε σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μόναχα να απαντήσω θα ήθελα για το... να έχω απαντήσεις για το ερώτημα που απίφθηνα στον κύριο Κολούτσι και στους άλλους. Ο αθλητισμός δεν βρίσκεται τώρα μέσα στην ε, πολιτική της Ευρώπης για το 2020 και η εκπαίδευση είναι φυσικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως θα μπορούσαμε ίσως να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική αθλητισμού και με επίσημο τρόπο να περιληφθεί στη στρατηγική του, της Ευρώπης 2020. Νέοι αθλητές, καταπολέμηση του ντόπινγκ και άλλα θέματα που είναι επίκαιρα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ενταχθούν στις οριζόντιες πολιτικές της Ευρώπης 2020. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για λεπτομέρειες αλλά περισσότερο για οριζόντιες πολιτικές. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η μέρημνα να γίνει κομμάτι της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Πόλγκερ και πάλι και μετά οι εμπειρογνώμονες εάν θέλουν να προσθέσουν κάτι ή αν θέλουν να σχολιάσουν και να κάνουν νέες προτάσεις μετά από αυτά που ακούσα. Ο κ. Πόλγερ έχει το λόγο και πάλι. Θα πάρετε το λόγο αργότερα οι υπόλοιποι. Πόλγερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να μου επιτρέψετε να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Για τη χρηματοδότηση. Εκ νέου και τον ερασιτεχνικό ή λαϊκό μάλλον αθλητισμό. Συμφωνούμε για τη σημασία που έχει ο λαϊκός αθλητισμός και θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα οποία μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αντικαταστήσει τις τοπικές αρχές για να νοικοδομηθούν ας πούμε τα τοπικά ποδοσφαιρικά σωματεία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρηματοδοτήσουμε τις διασυνοριακές δραστηριότητες τις οποίες ε, εμπλέκονται οι ε, οργανώσεις αυτές, η ανταλλαγή χρηστών πρακτικών, Σύντομα θα ανακοινώσουμε τα προγράμματα που θα υποστηριχθούν φέτος και τις προπαρασκευαστικές δράσεις για τον αθλητισμό θα υπάρξουν 12 προγράμματα που θα στηριχθούν χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον τομέα του ντόπινγκ και της καταπολέμησης του κοινωνικού ακοπλισμού μέσω του αθλητισμού. Αυτό προσθέτει μια διαφορετική έποψη θα έλεγα στα θέματα και του εθελοντισμού στον αθλητισμό, που και αυτό είναι κάτι που αφορά τον λεγόμενο λαϊκό αθλητισμό. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν λοιπόν και προτείνουμε να τα κάνουμε σε ένα μελλοντικό αθλητικό πρόγραμμα. Γύρω από το mainstreaming πράγματι θα υπάρξει ένα κενό στη χρηματοδότηση των αθλημάτων το 12 και το 13. Γι' αυτό κάνουμε μια έντονη προσπάθεια να εντάξουμε τον αθλητισμό σε άλλους τομείς. Ξεκινάμε με τα προγράμματα για την νεότητα. Θα προτείνουμε στις αρμόδιες διαχειριστικές επιτροπές ε, των προγραμμάτων που αφορούν την νεότητα να συμπεριλάβουν τον αθλητισμό σαν ετήσια προτεραιότητα για το 12 και το 2013. Αυτό είναι ένα παράδειγμα mainstreaming. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι δαπανώνται αρκετά χρήματα σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τον αθλητισμό, ιδιαίτερα για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Αυτό είναι βασικό θέμα, λιώδες θα έλεγα επιστημονικό, γιατί εφευρίσκονται και αναπτύσσονται συνεχώς νέες μέθοδοι για τον ντόπινγκ, νέες ουσίες, και πρέπει να δημιουργούνται και νέες μέθοδοι ανείχνευσης. Συνεπώς τα προγράμματα τα ερευνητικά σαφώς και συνεισφέρουν ε, στην επιστημονική αυτή δουλειά. Υπάρχουν επίσης ερωτήσεις για τον λεγόμενο εραστεχνικό αθλητισμό και την ερμηνεία που δίδεται για την κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με τον αθλητισμό και την ανάγκη για νομική ασφάλεια και βεβαιότητα. Όταν υιοθετηθεί η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνοδεύεται από ένα έγγραφο εργασίας το οποίο θα καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου, του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και της νομολογίας έτσι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν και θα μπορέσουν να προβλέψουν, θα έλεγα, την εξέλιξη των προγραμμάτων. Θα έχουμε ένα μεγαλύτερο, υψηλότερο ποσοστό προβλεψιμότητας. Αυτό αφορά κυρίως τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Μέχρι τώρα οι κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις είχαν σαν στόχο πιο πολύ τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ξέρουμε ταυτόχρονα ότι η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών είναι μία από τις τέσσερις βασικές αρχές της αρχικής συνθήκης της Ένωσης, της συνθήκης της Ρώμης. Αυτό εφαρμόζεται λοιπόν και στους ε, ρασιτέχνες αθλητές. Όταν μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη για επαγγελματικούς σαν παράδειγμα λόγους και ασκούν ένα άθλημα, θέλουν να συνεχίσουν να ασκούν αυτό το άθλημα στην καινούργια χώρα υποδοχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν εμπόδια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι συμβατό με, τις, με τη βασική αρχή της ελεύθερης διακίνησης. Ολοκληρώνουμε σύντομα μια μελέτη γύρω από την εφαρμογή των περιορισμών εθνικότητας στον τομέα των αθλητικών και ελπίζουμε αυτό να βοηθήσει να προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα και να είναι πιο εύκολο για μας τους πολίτες όταν ασκούμε το δικαίωμα μετακίνησης να έχουμε και το δικαίωμα άσκησης της αθλητικής δραστηριότητας που επιθυμούμε. Μια άλλη ερώτηση είναι το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερο κόσμο στον αθλητισμό και πόσο θα συμπεριλάβουμε τον αθλητισμό στις προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Συνδέονται τα δύο αυτά θέματα. Μέσω της ΧΕΤΑ. ΧΕΤΑ σημαίνει στα αγγλικά ε, γυμναστικές δραστηριότητες που βελτιώνουν την υγεία. Να πείσουμε λοιπόν όλο και περισσότερο κόσμο να ασκείται αυτό όχι μόνο προς προσωπική είναι ευχαρίστηση αλλά όσο περισσότεροι αθλούνται και ασκούνται τόσο περισσότερο υγιείς θα είναι, θα λείπουν λιγότερα από τη δουλειά τους, θα εργάζονται καλύτερα, θα είναι ευτυχέστεροι και αυτό θα βοηθήσει τους στόχους αηφόρου ανάπτυξης και απασχόλησης για το 2020 και σε της άλλης επειδή θα είναι υγιέστερος ο κόσμος μειώνεται και το κόστος των ασθενειών στα πλαίσια των συστημάτων πρόνοιας. Ταχέτα λοιπόν οι ε, γυμναστικές δραστηριότητες και ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν και οικονομικά θετικά με σοβαρό τρόπο. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω. για τις προτεραιότητες της κυρίας Χόνιμπολ. Η ανακοίνωση θα καλύπτει θέματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα προτείνουμε την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό και αναφερόμαστε και στο δικό σας ψήφισμα, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα ακολουθήσει την έκδοση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η δική σας, το δικό σας ψήφισμα θα καθορίζει ορθότερα και πιο συγκεκριμένα τις προτεραιότητες μας για το μέλλον. Δεν δόθηκε απάντηση νομίζω στο ερώτημα για τον προπολογισμό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δώσετε μια απάντηση για το θέμα αυτό. Αμικρόφωνος ο της Κομισιόν. Νομίζω ότι ο κύριος Λόκεργατ αναφερόταν στα προπαρασκευαστικές δράσεις. Γιατί αυτά είναι τα μόνα χρήματα τα οποία μπορούμε να οραματιστούμε προς το παρόν. Πρόκειται για 3 εκατομμύρια συν τα ποσά για τα ειδικά γεγονότα, τα έκτακτα γεγονότα. 7 εκατομμύρια συνολικά έχουν εγγραφεί από το Ευρωπαϊκό Προπολογισμό στον προπολογισμό, ο οποίο δεν ενεκρίθη. Λοιπόν, α ελπίσουμε ότι θα επιβιώσει και αυτή η γραμμή του προπολογισμού για το 2011 στι διαπραγματεύσει που πρέπει να λάβουν τώρα χώρα. Και το άλλο ερώτημα το οποίο τέθη. Ναι, ναι, η συμμετοχή των εμπλεκομένων. Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει κάτι τέτοιο. Η Κομισιόν οργανώνει, οργανώνει κάθε χρόνο το λεγόμενο αθλητικό φόρουμ. το φόρουμ αυτό ασχολείται με επίκαιρα θέματα και προσκαλούνται όλοι οι αθλητικοί φορείς, μεγάλοι, μεσαίοι και μικροί. Προσκαλούνται και οι ευρωβουλευτές, λοιπόν, είναι ένα σημαντικό γεγονός. Το επόμενο, θα γίνει, επόμενο, το επόμενο φόρουμ θα γίνει στη Βουδαπέστη στο τέλος του Φεβρουαρίου. Ελπίζουμε ότι πολλοί από εσάς θα μπορείτε να είστε παρόντες εκεί. Αυτό είναι και μια πρωτοβουλία της Ουγγρικής Προεδρίας ότι αυτή τη φορά θα γίνει αμέσως μετά από την άτυπη συνεδρία των Υπουργών Αθλητισμού μάλλον αμέσω πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Αθλητισμού. Επομένω, τα πορίσματα του φόρουμ μπορεί να πληροφορήσουν καλύτερα και του Υπουργού Αθλητισμού. Είναι λοιπόν μια ευρεία συνάθρηση και συγκέντρωση των εμπλεκομένων στο αθλητικό φόρουμ. Και υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα συμμετοχή των αθλητικών φορέων, αυτά που γίνονται από το Συμβούλιο. Σήμερα το απόγευμα η Βελική Προεδρία θα θέσει μια πρόταση για έγκριση, μια απόφαση η οποία θεσπίζει ένα διαρθρωμένο διάλογο με τις αθλητικές οργανώσεις. Δεν είναι μονάχα μπλα μπλα μπλα. Δημιουργεί λοιπόν το πλαίσιο για συνεχή διάλογο μεταξύ αθλητικών οργανώσεων και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανόμενου. Αλλά πέραν αυτών έχουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση η Κομισιόν επαφές με ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους στα θέματα αυτά. Εγώ είχα πάει στην Ολυμπιακή Επιτροπή για να συναντήσω τους εμπλεκομένους στον τομέα αυτό χθε. Πέρα λοιπόν αυτών των γεγονότων οροσύμων υπάρχει η καθημερινή μας δραστηριότητα που συνεχίζεται αενάως. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Κολούτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω το τελευταίο. Θέλω να γίνει μια διάκριση μεταξύ εραστεχνών και επαγγελματιών. Κάποιος παραπονέθηκε πως μετά την θέση ενισχύ της συνθήκης δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα του αθλητισμού όπως το ντόπινγκ ε, κτλ. Μην ξεχνάτε πως οι εμπλεκόμενοι δεν έχει σημασία ποιοι είναι το άθλημα που εκπροσωπούν. Έχουν μια πλατφόρμα να συζητούν τα πάντα. Και αυτή η πλατφόρμα λέγεται κοινωνικός διάλογος. Κοινωνικός διάλογος. Όταν είπα στην αρχή σήμερα το πρωί πως ο αθλητισμός παραμένει ευθύνη των εμπλεκομένων, παραμένει εάν αυτοί το θελήσουν, έχουν ένα μέσο ε, να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν, η Ένωση παίζει ένα ρόλο. Ποιο ρόλο? Να προωθήσει τον διάλογο. Ο διάλογος αυτός είναι μια ευκαιρία. Εγώ δεν μπορώ να αναγκάσω κανέναν εδώ πέρα να κάνει διάλογο αν δεν το θέλει και αν δεν του αρέσει ο άλλος. Α, τουλάχιστον μπορώ να σας φέρω εδώ και να συζητήσουμε και ίσως τελικά να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Γιατί να κατηγορούμε συνέχεια κάποιον άλλον, ένα πρόσωπο, ένα θεσμικό όργανο, εάν κάτι δεν δουλεύει. Έχουν μέσο να το κάνουν. Ο κοινωνικός διάλογος έχει επίσης και ένα άλλο όφελος. Η εντύπωση που έχουμε όλοι είναι πως κάποιοι εμπλεκόμενοι στον αθλητισμό προσωπούνται περισσότερο από άλλους. Γεγονός. Κάτι θετικό του κοινωνικού διαλόγου, καθώς ε, πρόκειται για διάλογο μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, είναι το εξή. Σε κάποιους τομείς δεν υπάρχουν εκπρόσωποι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Π.χ. στο ποδόσφαιρο, ο κοινωνικός διάλογος είχε το αποτέλεσμα να αναγκαστούν τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη να δημιουργήσουν έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Και προσπαθούν τώρα να κάνουν ένα κοινωνικό διάλογο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα άλλα αθλήματα. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, ε, Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω τίποτα εγώ για τον προϋπολογισμό Η γυναίκα μου τα κανονίζει τα οικονομικά. Ας υποθέσουμε πως έρχεται η γυναίκα μου και μου λέει «Μικέλε, χρειαζόμαστε ένα εκατομμύριο να αγοράσουμε αυτό το σπίτι». Λέω, θα της πω «Ε, Λίσμπετ, δεν γίνεται, δεν έχουμε λεφτά». Αλλά ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να πάρουμε ένα μικρότερο σπίτι. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή από κάτι συγκεκριμένο. Πόσο κοστίζει μια ευρωπαϊκή εκδήλωση. Σταματάω εδώ. Αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τα προβλήματα του προϋπολογισμού, την έλλειψη κονδυλίων, επομένως μπορείτε να καταλάβετε ότι για μας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό και ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια κονδύλια. Όσα και να έχουμε, δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα σπίτι ενός εκατομμυρίου. Ο κύριος Κέρκεμπι έχει το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση τι μπορείτε να κάνετε για μας εδώ εκπροσωπώντας οργανώσεις των λαϊκών αθλημάτων. Εμείς δίνουμε μια σταθμισμένη προσοχή θα έλεγα στον λαϊκό αθλητισμό, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και γενικότερα στην αθλητική δραστηριότητα και τη γυμναστική δραστηριότητα. Η τηλεόραση αν τη βλέπετε το μόνο που δείχνει είναι τα ανταγωνιστικά αθλήματα, ποδόσφαιρο κτλ. Προκαλεί όμως πολιτικό ενδιαφέρον το τι ε, θέλουν και τι ενδιαφέρει την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθηγητής Βλαντιμίρ Αντρέ αναγνωρίζει ότι είναι πρόβλημα να συνεχίσουμε να παραπέμπουμε σε ένα μοντέλο το οποίο αποκλείει τα δύο τρίτα της πραγματικότητας. Τα δύο τρίτα που δεν ανήκουν σε ένα σύλλογο, που δεν ανήκουν σε ένα σωματείο, που δεν ενδιαφέρονται να είναι οι καλύτεροι. Είμαστε στη διάθεσή σας για ιδέες. Κάποιες από τις ιδέες που ακούστηκαν για το Εράσμος πρέπει να αναπτυχθούν. Οργανώνουμε 40 με 100 χιλιάδες ε, γεγονότα αθλητικά σε όλη την Ευρώπη σε ετήσια βάση. Είναι κάτι το αβίαστο, το εύκολο και έτσι ακούγεται και η φωνή όλων των Ευρωπαίων. 100 εκατομμύρια θα πρέπει να είναι ο στόχος Ευρωπαίων που αθλούνται και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει όραμα να βοηθήσει αυτούς που έχουν αναπτυξιακό δυναμικό στη διάθεσή τους και να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πιστεύω και εγώ πράγματι ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε το διάλογο, να κρατήσουμε το διάλογο ζωντανό μεταξύ αθλητικών ενώσεων και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό κάνουμε. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα διαλόγου. Ο διάλογος υπάρχει. Προφανές όμως είναι ότι για μας σε ό,τι αφορά τους πόρους είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει μια συνθήκη και ένα νέο άρθρο στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό. Τον αθλητισμός γίνεται αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της ότι θα πρέπει από την αρχή να γίνει κάτι έστω και αν έχει συμβολικό χαρακτήρα στο να υπάρχουν πόροι διαθεσμοί για αυτή την κατηγορία για τον αθλητισμό για τα ομαδικά αθλήματα στην Ευρώπη. Εμείς δεν ζητούμε πόρους. Ζητούμε όμως το σεβασμό της αυτονομίας μας σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα λήψης απόφασης για την αυτοδιοίκηση του αθλητισμού. <clears throat> Χάρη στο μοντέλο πυραμίδας καταφέραμε να χρηματοδοτήσουμε και τον αθλητισμό στη βάση και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν στο μέλλον είναι να μας ακούτε και να έχετε συνεχή διάλογο μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Ο Πάντρικ έχει το λόγο. Για να... Ευχαριστώ για να ολοκληρώσω. Συμφωνώ με τον συναδελφό που μίλησε για την αυτονομία του αθλητισμού και πρέπει να μείνουν απ' έξω οι πολιτικοί. Δεύτερον, είναι λυπηρό να ακούμε σήμερα πως με την εφαρμογή του άρθρου 165 από ό,τι άκουσα δεν θα υπάρχει πρόγραμμα μέχρι το 2015 και μετά λυπηρό και δεν θα χαρούν πολύ και οι πολίτες της Ευρώπης και τέλος κάτι θετικό χαρικά που άκουσα τον συνάδελφο από την Ουγγαρία για τα της Ουγγρικής Προεδρίας και για το πόσο δραστηριοποιούνται στον τομέα του ε, αθλητισμού και είναι θετικό αυτό και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στη Βελγική Προεδρία, η κυρία Φερμέρης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, Πρώτα απ' όλα ο υπουργό μου, ο κύριο Μέτερ, ο φλαμανδό υπουργό αθλητισμού, είχε μία άλλη συνεδρίαση. Προετοιμάζει το Συμβούλιο δηλαδή, γι' αυτό δεν μπορεί να παραστεί. Οπότε θα σας ενημερώσω πως ε, ελπίζω το Συμβούλιο το απόγευμα να είναι κάτι παραπάνω από μπλε μπλα μπορούμε να πούμε πως είναι μια ιστορική συνάντηση από την έννοια πως για πρώτη φορά συναντώνται στο Συμβούλιο οι Υπουργοί Αθλητισμού. Γιατί ξέρετε αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προσθέσει τη λέξη αθλητισμό στο Συμβούλιο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εκπαίδευσης πολιτισμού και αθλητισμού. Και αυτό είναι ένα πρώτο μήνυμα Εντό του Συμβουλίου και θα συνεχίσουμε βεβαίω να εργαζόμαστε στον τομέα του αθλητισμού. Για τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι ο δομμένος διάλογος με τον τομέα του αθλητισμού, κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού και καταπολέμηση του ντόπινγκ. Για τον δομμένο διάλογο ξέρετε πως δίνουμε προτεραιότητα σε συζητήσεις ε, που έχουν ξεκινήσει επί Ισπανικής Προεδρίας και τις συνεχίζουμε. Προσπαθούμε να βρούμε διάφορους ε, μηχανισμούς και να δούμε και ποιοι είναι οι υπάρχοντες μηχανισμοί, ειδικά το φόρουμ το οποίο οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης ανέφερε ο πρόσωπος της Κομισιόν πως ε, απόψε το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με ένα ψήφισμα για το δομημένο διάλογο όπου σκοπεύουμε να θέσουμε ένα πλαίσιο διαλόγου και ειδικά να υπάρξει ένα στοιχείο υψηλού επίπεδου σε αυτούς τους μηχανισμούς θα μπορέσουμε έτσι στο περιθώριο του Συμβουλίου να έχουμε και μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων και πρόθεσή μας είναι όπως είπα πρώτα απ' όλα να καταστεί σαφές αυτό το πλαίσιο και μετά να οδηγηθούμε σε μια πρώτη έτσι, συνάντηση, ίσως τον Δεκέμβριο, ακόμα επί Βελγικής Προεδρίας. Η δεύτερη προτεραιότητά μας για τη Βελγική Προεδρία, για την κοινωνική ένταξη στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού είναι πως θα βγάλουμε συμπεράσματα για το ρόλο του αθλητισμού ως πηγή και κινητήρα κοινωνικής ένταξης ε, ως ένα σημαντικό μήνυμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής μέσω του αθλητισμού. Και βεβαίως ε, αυτό ε, ταιριάζει και με μια, ένα συνέδριο ειδικών που έχει οργανωθεί επί Βελικής Προεδρίας και θέλουν οπωσδήποτε οι Υπουργοί να το δουν με βάση την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για να δούμε τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο θέμα, ντόπινγκ και καταπολέμησή του, είναι σημαντικό. Και εδώ πέρα προετοιμάζουμε συμπεράσματα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή καταπολέμηση του ντόπινγκ. Τονίζουν τα συμπεράσματα αυτά τη σημασία συντονισμού, Ένωσης και κρατών μελών, ειδικά όσον αφορά τη συνεδρία στη Γουάντα. Σκοπεύουμε με τα συμπεράσματα αυτά να ενισχύσουμε το ρόλο της Ένωσης και της Ευρώπης συνολικά για να αντιμετωπίσουμε τον τόπινγκ. Επίσης, το ανέφερε και η κυρία Μποσκούρτ και ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν για την εκπροσώπηση δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γουάντα. Είχαμε κάποιε άτυπε συζητήσει στο επίπεδο των Υπουργών και βεβαίω θα συνεχιστούν αυτά και επί της Προεδρής μας. Επίσης, Υπάρχουν δύο άλλα σημαντικά σημεία, το θέμα των ε, εθελοντών και η εκπαίδευση και κατάρτιση ε, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί στο πλαίσιο του EQF, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και μέσα Δεκεμβρίου θα γίνει μια διάσκεψη ειδικών η Ευρωπαϊκή ημέρα των εκπαιδευτών όπου είστε προσκεκλημένοι εάν θέλετε. Οπότε σας παρουσίασα τις προτεραιότητες μας και ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου πως η Βελγική Προεδρία θα καταβάλει μια πρώτη προσπάθεια για να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική του αθλητισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε φτάσει στο τέλος της ακρόασής μας. Μια ακρόαση η οποία ήταν ιδιαίτερα επίκαιρη, ιδιαίτερα σημαντική ήταν ακριβώς την κατάλληλη χρονική στιγμή όπως είπα προηγουμένως. Θέλω να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου στους εμπειρογρόμονες που ήρθαν εδώ. Συγγνώμη που ήμουν πολλές φορές πολύ αυστηρή μαζί σας για τη χρήση του χρόνου, αλλά αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τηρήσουμε το χρονοδιαγράμμα. Κάποιον νομίζω ότι τον ε, περιέκοψα στη χρήση του λόγου, ελπίζω να με συγχωρήσει και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και μια πολύ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα πρέπει να δείξει μια μεγαλύτερη δημιουργικότητα και μεγαλύτερη φαντασία για τα θέματα αυτά για να μπορέσει να γίνει πλήρης εφαρμογή του άρθρου 165. Έχουμε φυσικά την δυνατότητα του mainstreaming σε πολλούς άλλους τομείς. Αλλά πρέπει να υπάρξει και μια συνειδητοποίηση της ανάγκης συντονισμού. Θα πρέπει να υπάρξει και η πολιτική ε, θέληση και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πόλγκερ από την Κομισιόν και ελπίζω ότι ο ενθουσιασμός που έχετε ε, δείξει θα εφαρμοστεί και στον τομέα αυτό. Ένα ακόμα πράγμα θέλω να κάνω είναι σήμερα κάτι το, έγινε σήμερα κάτι το οποίο πρέπει να πω ανοιχτά ότι με τρόμαξε ότι αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα του επιστητού. Δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθο όπω κάναμε και στη στρατηγική Λισαβόνα. Να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και στο τέλο να μην γίνει τίποτα. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ευρύτατο το υπόβαθρο του αθλητισμού και αυτό το υπογράμμισαν και οι εμπειρογνωμονέ μα. Αυτό μπορεί να το τονίσει κανεί σε επίπεδο εισαγωγικό. Αλλά σα παρακαλώ, α εστιάσουμε την προσοχή μα σε λίγα μονάχα θέματα τα οποία μπορούμε να τα φέρουμε σε υλοποίηση στα επόμενα χρόνια. Αν έχουμε τέσσερα ή πέντε σημεία τα οποία εμεί μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αυτό θα είναι πιο επωφελέ. Θέλω να πω επίση και κάτι ακόμα. Έχουμε δύο συγκεκριμένα καθήκοντα αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, να υποστηρίξουμε αυτό το οποίο θέλουμε όλοι, δηλαδή ώστε το περισσότεροι άνθρωποι να ασκούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικέ δραστηριότητε να βοηθούν λοιπόν ως ε, μέλη ραστεχνικών συλλόγων και ως οπαδοί. Και αυτό είναι και ένας τρόπος επίσης να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό, να τονίσουμε ότι μέσα στα πλαίσια του έτους εκπαίδευσης και αθλητισμού να παίξουμε ένα μεγάλο ρόλο. Αλλά έχουμε και ένα δεύτερο καθήκον για τον επαγγελματικό αθλητισμό, να βοηθήσουμε τον επαγγελματικό αθλητισμό ώστε όλοι αυτοί μας θέτουν ερωτήμα παραγωγή για τους μάνατζερ των παικτών, τους player agents και άλλα τεχνικά θέματα που έχουν να κάνουν με τον επαγγελματισμό στον αθλητισμό να επιληθούν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί οργανώσεις όπως η UEFA έχουν τη δυνατότητα μονάχα ένα μέρος αυτών των προβλημάτων να αντιμετωπίσουν και ίσως υπάρχει δυνατότητα εμείς από κοινού με τις επαγγελματικές αθλητικές οργανώσεις να βρούμε τρόπο και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες δράσης και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ήδη υπάρχοντα εργαλεία για να προχωρήσουμε. Θέλω να σας υπενθυμίσω εξάλλου ότι στην πραγματικότητα όλες αυτές οι δραστηριότητες ξεκινήσανε με την υπόθεση Μπόσμαν στη δεκαετία του 1990. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ουσιαστικά αντιμετωπιστεί από τους Ευρωπαίους βουλευτές το θέμα του αθλητισμού. Αλλά έκτοτε υπήρξε μια συνειδητοποίηση ότι πρέπει να υπάρξει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και δεν μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα του αθλητισμού σαν είναι μονάχα ζητήματα ανταγωνισμού. Και αυτό συνέπτεται με αυτό που είπατε προηγουμένω για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αθλητισμού. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε ότι εμεί θα επηρεάσουμε και θα περιορίσουμε την αυτονομία σα. Ο τότε Πρωθυπουργό Κόλ είχε εξασφαλίσει να υπάρχει η αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων. Αλλά από τη δική μας πλευρά εμείς θέλουμε να δούμε αν μπορούμε μαζί με την Κομισιόν να κάνουμε κάτι μαζί και χαίρομαι που η Βελική Προεδρία έχει δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτόν τον τομέα και θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε και τη δική σας άποψη μαζί με την Κομισιόν για το αν μπορούμε να κάνουμε κάτι στο μέλλον για να διευκολύνουμε και την δουλειά των αθλητικών οργανώσεων. Και τώρα μην έχουμε προγράμματα για το 2012 και το 2013 δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε τίποτα στον τομέα αυτό. Κρίμα που έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά έτσι είναι και γι' αυτό δεν πρέπει εμείς να απογοητευόμαστε, θα πρέπει να ενισχύσουμε την Επιτροπή να μας παρουσιάσει τις ιδέες της και να την υποστηρίξουμε για να τις εφαρμόσει, να βρούμε άλλους δρόμους για να επιτύχουμε τα αποτελέσματα αυτά και μετά όλα αυτά τα οποία θέλουμε εμείς να μπορέσουν να υλοποιηθούν σε ειδικά γεγονότα, σε προπαρασκευαστικές δράσεις, ώστε να καταλάβουν οι πολίτες ότι ναι, ακόμα γίνεται κάτι στον τομέα του αθλητισμού, μπορούμε να δράσουμε και να υπάρξει αυτή η υποστήριξη. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους σας και αν ήμουν κάποτε αυστηρή με τον κύριο Κέλλη και άλλους, νομίζω ότι ίσως δεν συμφωνείτε με την άποψή μου για την γραπτή δήλωση για μένα είναι σημαντικό να, <laughs> να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση. Λοιπόν, να αφήσουμε κατά μέρο τη γραπτή δήλωση. Κλείνω την ε, ακρόαση και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αφήσετε την αίθουσα γιατί πρέπει να κάνουμε συνεδρίαση των συντονιστών και ευχαριστώ και τους διερμηνείς.